Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω πως ε, ήδη πέρασαν τα πέντε λεπτά ανοχής και επομένως θα πρέπει να ξεκινήσουμε ε, διότι έτσι όπως μας είχε ήδη προειδοποιήσει ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς θα είναι μαζί μας μέχρι τις 8 και Ξεκινάω αμέσως με το πρώτο σημείο της ημερησίας διατάξεως που αφορά την έγκριση της ημερησίας διατάξεως. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, το προσχέδιο εγκρίνεται χωρίς καμία τροποποίηση. Όσον αφορά τις ανακοινώσεις του Προέδρου, μπορώ να σας πω το εξής. Η διερμηνία ε, ε, ε, θα είναι διαθέσιμη σε 20 γλώσσες, χωρίς λετωνικά, εστονικά και μαλτέζικα. Ως συνήθως η συνεδρίαση θα είναι web-streamed. Περνάω αμέσως στο δεύτερο σημείο, που είναι βεβαίως το κυρίως θέμα ε, τη σημερινής μας ημερήσιας διάταξη και συνάντηση είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον Φραν Τίμερμαν, Τίμερμαν πρώτο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, ο οποίος ε, ασχολείται με την καλύτερη νομοθέτηση, της διαθεσμικές σχέσεις, καθώς επίσης ασχολείται και με την βιωσιμότητα και την αηφορία. Ως πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι σε θέση επίσης να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις όσον αφορά την οργάνωση λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον αντιπρόεδρο ε, Φρανς Τίμερμανς και ε, θα ε, οργανώσουμε δύο γύρους ερωτήσεων ως ήθιστε. Πρώτα θα ακούσουμε το, την εισαγωγική ομιλία του ε, κυρίου Αντιπροέδρου, καμιά δεκαριά λεπτά και μετά ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων από πλευρά των συντονιστών των πολιτικών ομάδων και μετά δεύτερο γύρο ερωτήσεων από τους συναδέλφους της ε, δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Ε, ο ΔΕ Αντιπρόεδρος θα απαντήσει αν μπλόκο στις ερωτήσεις ε, κάθε φορά. Του δίνω αμέσως το λόγο για την εισαγωγική του παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Έχω πολλά πράγματα να πω σήμερα. Θα τα πω όμως στα αγγλικά. Καλό απόγευμα ή μάλλον καλό βράδυ κυρίες και κύριοι. Όντως, ε, στο χαρτοφυλάκιό μου έχω πολλά ε, θέματα και υποχρεώσεις. Ε, και επομένως ενώπιον του Κοινοβουλίου ε, πρέπει να πω και μετά μάλλον από αίτημα του Κοινοβουλίου προστέθηκε στο χαρτοφυλάκιο και η βιώσιμη ανάπτυξη και σας είμαι ιδιαίτερος ευγνώμων για την προσθήκη αυτή γιατί πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έρχεται και κουμπώνει πάρα πολύ καλά με όλα τα υπόλοιπα θέματα τα οποία είχα ήδη στο χαρτοφυλάκιό μου. Η βιωσιμότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί σωστά εάν η προσέγγιση είναι συνολική ένα από τα συμπεράσματα στα οποία μπορώ ε, να φτάσω μετά από 100 μέρες σε αυτή τη θέση είναι ότι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση άσχετα από το θεσμικό όργανο που εκπροσωπεί κανείς ε, δουλεύουμε συνήθως ε, σε κενά και σε φυλάκους και αυτό δεν είναι δυνατόν να το δεχτούμε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε δουλεύοντας σε συνεργασία και σε κύκλους όπου ε, και η κοινωνική ανάπτυξη θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται οπωσδήποτε την ε, ε, ανάπτυξη, στη βιώσιμη ανάπτυξη. Χωρίς αυτήν η βιώσιμη ανάπτυξη δυστυχώς δεν είναι δυνατόν να είναι επιτυχής. Ε, είμαι απολύτως πεπισμένος ότι θα πρέπει να ενταχθούν μια σειρά πολιτικών από την οπτική γωνία της βιώσιμης ανάπτυξης και ότι θα πρέπει να εξυπηρεθούν συνέργειες από διάφορες οπτικές γωνίες έτσι ώστε να έχουμε επιτυχή αποτελέσματα. Εγώ βλέπω τον ρόλο μου στην Κομισιόν σαν πρώτο αντιπρόεδρο όχι σαν κάποιο που θα πρέπει ε, να κάνει τη δουλειά ενός επιτρόπου που θα είναι ε, ε, που θα ελέγχει τον κάθε επίτροπο αν κάνει καλά τη δουλειά του αλλά ότι θα, θα υπάρχει μια σωστή συνέργεια ανάμεσα στους διαφόρους επιτρόπους και τα διάφορα χαρτοφυλάκια δηλαδή αυτός που είναι υπεύθυνο για το περιβάλλον να μπορεί να συνεργάζεται με αυτό που είναι υπεύθυνη για κοινωνικά θέματα. Η κυκλική οικονομία επίσης ε, είναι πάρα πολύ σημαντική, κυρίως τώρα στα πλαίσια της συζήτησης του προγράμματος ε, ε, Juncker και γι' αυτό ακριβώς συνεργάζομαι και με τον Επιτροπο Κατάινεν και με τον, σήμερα το πρωί μίλησα και με τον Επιτροπο Μουέντερ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε όλα τα στοιχεία τα οποία εκπροσωπούν μέσω των χαρτοφυλακίων του οι Επίτροποι και να συνδράμουμε όλοι στην άπτυξη του, του προγράμματος Juncker. Πριν ε, ε, αναφερθώ σε όλα τα ζητήματα, θα ήθελα να πω ότι το κυριότερο θέμα το οποίο θέλω να θίξω είναι να σας πω το εξής. Εάν μπορέσουμε ε, να φτάσουμε σε συμφωνία σχετικά με το ποιοι είναι οι στόχοι μας και ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς χωρίς να τίθενται να αμφιβόλο και να αμφισβητούνται οι στόχοι αυτοί ήδη θα έχουμε κάνει ένα πάρα πολύ καλό βήμα. Έτσι θα πρέπει να καθορίσουμε την ε, ημερήσια διάταξη των εργασιών μας. Ε, ξέρω ότι η καλή νομοθέτηση, η σωστή, ε, ε, η σωστή νομοθετική αντιμετώπιση είναι κάτι πάρα πολύ καλό και κάτι πάρα πολύ θετικό. Ξέρω στα παρελθόντα ότι υπήρχαν προβλήματα όσον αφορά την απορρίθμιση, αλλά ε, ε, νομίζω ότι δεν αρκεί να θέτουμε στόχους. Το ζήτημα είναι η μεθοδολογία της επίτευξης των στόχων, να μην ε, θέτουμε σε αμφισβήτηση τους στόχους στο επίπεδο το οποίο θέλουμε να επιτύχουμε και να σας πω ότι εγώ αυτό που θέλω είναι ο κάθε ένας από τους επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της παρούσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι ε, ένας σε ο οποίος, ο θα ασχολείται με την ε, καλή ρύθμιση γιατί με τον τρόπο αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε μια συνολική αντιμετώπιση και σαν Επιτροπή να καταφέρουμε ε, να κάνουμε αυτό το βήμα προς την διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και προς την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα αλλά με τρόπο που το πέρασμα αυτό να μην είναι ούτε ασαφές από νομική άποψη, ούτε και βαρύ από άποψη οικονομική ή ε, γραφειοκρατική. Κατά αυτή την έννοια θα πρέπει τα θέματα να ε, αξιολογηθούν σωστά η καλύτερη ρύθμιση βεβαίως ε, συμπεριλαμβάνει και το ότι θα πρέπει να γίνεται μια μελέτη αντικτύπου όχι μόνο στην αρχή αλλά και σε όλη τη διάρκεια της νομοθετικής ε, διαδικασίας και να δούμε ότι εάν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στις προτάσεις της Κομισιόν να ξέρουμε ανα πάσα στιγμή ε, ποια μπορεί να, ποιος μπορεί να είναι ο αντίκτυπος στην πραγματική ζωή και ποιος μπορεί να είναι ο αντίκτυπος επί του αποτελέσματος. Θα πρέπει βεβαίως να να συζητήσουμε και τις διαθεσμικές συμφωνίες όσον αφορά την καλύτερη ε, νομοθεσία. Αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα. Είπα δύο λόγια λοιπόν όσον αφορά την ε, νέα δομή της Κομισιόν. Ε, θα ήθελα να υπογραμμίσω για μία ακόμα φορά ότι ρόλος του Αντιπροέδρου δεν είναι να τεκάρει ξανά και ξανά τους επιτρόπους, αλλά να διασφαλίσει την σωστή συνέχεια και συνεκτικότητα μεταξύ των πολιτικών και ότι ευθυγραμμίζονται η τα διάφορα μέτρα και αποφάσεις με, την, τον κεντρικό άξονα δράσεων του ε, Προέδρου Γιούγκερ και της Επιτροπής ε, Γιούγκερ. Δεύτερον, δεν, μας, ε, δεν θέλουμε να αμφισβητούν με τους στόχους, θέλουμε να δημιουργήσουμε το καλύτερο νομικό και νομοθετικό ρυθμιστικό περιβάλλον έτσι ώστε η επίτευξη των στόχων να γίνει με καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Θέλω να είμαι πολύ σύντομος γιατί ξέρω ότι οι ερωτήσεις θα είναι πολλές. Νομίζω ότι ξέρω μερικές από τις ερωτήσεις ε, που θα υποβληθούν. Ε, είναι, είναι βέβαιο ότι πρέπει να έχουμε αυτή τη δυνατότητα συζήτησης έτσι ώστε να αποσαφηνίζονται όλα τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε Τίμερ, μας λέει ο Πρόεδρος. Ε, ε μας κάνατε μια σύντομη εισαγωγική παρέμβαση έτσι ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο εμείς να σας υποβάλουμε ερωτήσεις. Θα δώσω πρώτα το λόγο στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και ξεκινώ με το ΕΛΚ και τον Πίτερ Λίζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής. Χαίρομαι που έχουμε σήμερα αυτή την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων. Νομίζω ότι θα πρέπει κατευθείαν όμως να ρωτήσω γιατί μας δίνεται αυτή η ευκαιρία τόσο αργά. Οι συντονιστές ε, ήδη στις 2 ε, Νοεμβρίου αποφάσισαν σχετικά με την βιωσιμότητα ότι θέλουμε να έχουμε μια συζήτηση μαζί σας και έχει περάσει πολλής χρόνος από τις 2 Νοεμβρίου μέχρι τις αρχές Μαρτίου και θα ήθελα να μπορούσα να καταλάβω γιατί χρειάστηκε να περάσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ε, η πρώτη θα έπρεπε να έρθει από εσά. Καλό θα ήταν να μπορούσαμε να συναντηθούμε και με την Επιτροπή Ήτρε από κοινού. Θα ήταν καλό να γίνει μια συνάντηση ε, με την Επιτροπή NB και Ήτρε. Και ο συντονιστή, ε, ε, προσπάθησαν οι συντονιστέ η Χριστιανή Κάρεν και οι συνεργάτε να οργανώσουν μια τέτοια συνάντηση. Ε, δεν ξέρω, θα ήθελα από εσά μια απάντηση. Γιατί χρειάστηκε τόσο πολύ χρόνο, ε, τι προβλήματα υπάρχουν σε αυτή την ε, κοινή συνάντηση. Όπως θα πούν και άλλοι συνάδελφοι, φαντάζομαι, και εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος με την απόσυρση του πακέτου σχετικά με τα απόβλητα θα ήθελα και προσωπικά θα ήθελα ε, να δω πώς μπορεί να ε, υπάρξει μια νέα πιο φιλόδοξη πρόταση σχετικά. Θα με ενδιαφέρει πολύ να ε, δω πώς θα είναι μια καινούρια πρόταση. Η ομάδα του ΕΛΚ αποδίδει μεγάλη σημασία αυτή στην νομοθεσία και δεν θα θέλαμε να παραβλέπουμε το ότι κάποια καλά μέτρα θα πρέπει να διατηρούνται. Παραδείγματο χάρη, ένα επίτροπο για το περιβάλλον προέρχεται από τη Μάλτα και στη Μάλτα ε, υπάρχουν διατάξει που δεν έχουν εφαρμοστεί και ακούμε τα τελευταία δύο-τρία χρόνια ότι όλο και κάτι θα αλλάξει, θα μεταφερθεί σε εθνικό δίκαιο η νομοθεσία, πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει. Όσον αφορά μια πιθανή αξιολόγηση των μέτρων, ε, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε την οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό και σχετικές προτάσεις για αποδυνάμωση αυτής της ε, οδηγίας. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να δείξουμε συνέπεια των πολιτών της Ευρώπης. θα πρέπει να δείξουμε όπως ε, στην περίπτωση με τους ε, κλασικούς λαμπτήρες ε, πυράκτωσης τι εναλλακτικά μέτρα υπάρχουν όταν προτείνουμε μια καινούργια οδηγία, μια απόσυρση κάποιων παλαιότερων μέτρων όπως να δείξουμε γιατί είναι καλύτεροι οι λαμπτήρες αλογόνου παραδείγματος χάρη να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις Ευχαριστώ Ματίας Γκρότερ, εκ των Σοσιαλιστών Ευχαριστώ πολύ Πολύ θετικό το ότι σήμερα μας δίνεται η ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής και στις ακροάσεις ε, προσπαθήσαμε εμείς το θέμα της βιωσιμότητας να το θέσουμε υψηλά στις προτεραιότητες. Ε, τώρα πέρασαν οι 100 ημέρες, το θέμα όντως της βιωσιμότητας όντως ε, έχει λάβει μεγάλη προσοχή και θέλουμε να ξέρουμε τώρα τι συμβαίνει. Ε, αποσύρθηκε το πακέτο για τα απόβλητα την περασμένη εβδομάδα νομίζω. Τώρα θα πρέπει να κοιτάξουμε προς τα μπρος, να δούμε ε, πώς προχωρούμε με την κυκλική οικονομία, πώς μπορούν οι προτάσεις να βελτιωθούν, πώς μπορούν να γίνονται καλύτερες ε, προτάσεις δεν θέλουμε απλώς να νομίζουμε ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση αναμονής όπου αναβάλλονται κάποια μέτρα. Θέλουμε να είμαστε θετικοί, να βλέπουμε θετικά το μέλλον, να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. και ελπίζω να μπορέσουμε το συντομότερο να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για να μπορούμε να αρχίσουμε ε, να δουλεύουμε και εδώ στο Κοινοβούλιο. Είχαμε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση ε, στην Επιτροπή, ήταν και ο Έντμος Στόιμπε ε, προσκεκλημένος και δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας με αντικείμενο την κατάργηση της γραφειοκρατίας. Έγιναν πολλές συζητήσεις με πολλές διαφωνίες και πολύ συχνά ξέρουμε ότι στα κράτη-μέλη δεν μεταφέρονται σε εθνικό δίκαιο σωστά οι διάφορες οδηγίες, οι διάφορες διατάξεις και πολλές φορές γίνεται και στρέβλωση των διατάξεων και θα θέλαμε από την Επιτροπή κάποια όθηση για να μπορέσουν να βελτιωθούν τα πράγματα. μερικές φορές η Επιτροπή είναι σαν ένα σάκος ε, τον χτυπάς και όλο και κάτι υπάρχει για να βγει από μέσα. Υπάρχουν διάφορα θέματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Οδηγία για τα είδα, τα 15 χρόνια και δεν έχει γίνει τίποτα και ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι είναι τόσα πολλά τα, τα 15 χρόνια και κάτι πρέπει να γίνει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τελικά οι διατάξεις οι οποίες ψηφίζονται να εφαρμόζονται στην πράξη, να μεταφέρονται σε εθνικό δίκαιο. Και τέλος θέλω να πω ότι Πολλές παρανοήσεις έχουν υπάρξει και ο Πέτερ ε, το ανέφερε ότι θέλαμε αυτή τη συνάντηση με την Ήτρε. Εμείς είμαστε βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, θέλουμε να υπάρχει μια ατμόσφαιρα συνεργασίας. Δεν είμαστε ε, εθνικό κοινοβούλιο. Αυτό το οποίο εμείς αποζητούμε είναι καλύτερη συνεργασία και αποφυγή των παρανοήσεων. Θέλουμε να συνομιλούμε για να αποφεύγουμε παρανοήσεις. Και το ότι έχουμε σήμερα αυτή τη συζήτηση είναι πολύ θετικό. Και οι διαφωνίες, που μπορεί και να μην υπάρξουν διαφωνίες, ε, καλό είναι να συζητούνται τα διάφορα θέματα και να ε, εξηγούνται όλες οι πτυχές των θεμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που σήμερα είστε μαζί μας. Ο συνάδελφος Πιέκα για τους ε, ε μεταρρυθμιστές και για το Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση και προ την Επιτρόπο Σεύκοβιτς ε, για την καλύτερη νομοθεσία είναι όμως το ερώτημα και γι' αυτό το θέτω σε εσά το ερώτημα. Βάση της σωστής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια συνθήκη οι συνθήκες μερικές φορές δεν είναι απόλυτα σαφείς. Μερικές φορές οι διατάξεις μας οδηγούν σε σχιζοφρενείς ερμηνείες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το, μείγμα, το ενεργειακό μείγμα. Αφενός μεν υπάρχει ε, η συνθήκη που δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευρείες δυνατότητες να δημιουργηθεί αυτό το ενεργειακό μείγμα. Από την άλλη πλευρά όμως λέγεται ότι δεν πρέπει να φύγονται τα δικαιώματα των κρατών μελών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιλέγουν τα κράτη-μέλη το ενεργειακό τους μείγμα. Και υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία όπου απαιτείται ομοφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όταν είναι διαφορετικές οι προτάσεις της Επιτροπής από τις προτάσεις των κρατών μελών. Δεν το έχει ξεπεράσει το πρόβλημα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. και στην νομοθεσία σχετικά με το εμπόριο εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος προέκυψε ένα σχετικό τέτοιο θέμα παρανόησης ή σχιζοφρενούς ερμηνείας. Μερικές φορές το γράμμα του νόμου, το γράμμα της οδηγίας είναι διαφορετικό από το πνεύμα της ε, μεταφοράς σε εθνικό δίκαιο. Τα κράτη-μέλη κάνουν διαφορετικές ερμηνείες. Απλώς χρησιμοποιούν τις προτάσεις ως βάση. οι ε, προτάσεις ε, για τον έλεγχο του ενεργειακού μείγματος στα κράτη-μέλη είπε ε, κάποιος συνάδελφος ότι θα πρέπει να ρυθμίζονται από τη συνθήκη. Θα μπορούσε όμως να ισχύει και το αντίστροφο. Ίσως θα έπρεπε τα κράτη-μέλη να έχουν περισσότερες αρμοδιότητες όσον αφορά τον καθορισμό του ενεργειακού μείγματος και να είναι υπεύθυνα τα κράτη-μέλη για, το βιώσιμο ενεργειακό μείγμα. Ποια είναι η δική σας γνώμη θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα γίνει κάποια αναθεώρηση αυτών των διατάξεων. Θα τηρήσουμε το γράμμα του νόμου ε, ώστε να μην υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες. Γιάννη Κέρτνα από τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Τίμερμανς. Όπως είπε ο Πίτερ Λίζε, αργήσατε να έρθετε να μας συναντήσετε εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ε, την έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ αναφέρεται αναφέρονται η κρίση για το νερό, της κλιματικής αλλαγής και της βιοποικιλότητας, Τρεις διαφορετικές κρίσεις, τρεις διαφορετικές απειλές για το περιβάλλον και την οικονομία. Σε μια άλλη έκθεση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ εξετάζονται οι μεγάλες τάσεις που θα επηρεάσουν τον κόσμο μέχρι το 2030 Ορισμένες από τις ε, σοβαρότερες απειλές που προβλέπονται είναι περιβαλλοντικής φύσεως και εκεί. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος επίσης στην έκθεσή της αναφέρει ότι η κλιματική αλλαγή και η έλλειψη και η μείωση της βιοποικιλότητας δημιουργούν σημαντικά μειονεκτήματα και αποτελούν μείζονες απειλές Εσείς αναφέρατε μερικά ωραία πράγματα για τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης κλπ. Αλλά αν δω την, το εργασία εργασίες της Κομισιόν και τις κατευθύνσεις αμέσως που παρουσίασε ο πρόεδρος Γιούνκερ διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν σημαντικά κενά στη δράση της Κομισιόν σε ό,τι αφορά το θέμα της ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Το κλίμα είναι μία από τις ε, δέκα προτεραιότητες σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όμως αυτό δεν έχει τόσο πολύ σχέση με τις απειλές όσο με την προμήθεια και τον φαντασμισμό ενέργειας. Οπότε ε, <clears throat> εκεί υπάρχει κενό και λέτε ότι μας ευχαριστείτε που έχουμε καθορίσει ως βασική προτεραιότητα τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οπότε αυτό με οδηγεί σε δύο ερωτήσεις. Δεδομένης της σημασίας της βιώσιμης ανάπτυξης τόσο για το περιβάλλον όσο και για ε, την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα, για το μέλλον όλων μας, η ομάδα μου και πιστεύω ένα μεγάλο τμήμα της Επιτροπής αυτής θα ήθελε θα ήθελα να σας ζητήσουν να μας εκθέσετε το όραμά σας για αυτά τα θέματα. Πότε μπορούμε να περιμένουμε κάτι τέτοιο. Μετά, για το θέμα της βιοπικιλότητας, την οποία πολλοί ονομάζουν η σιωπηρή κρίση. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπίζουμε. Το αναφέραμε αυτό και στην έκθεσή μας. Είχαμε την ανασκόπηση της ε, στρατηγικής ε, βιοπικιλότητας τη Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν δείτε αυτή και την έκθεση για την κατάσταση περιβάλλοντος θα διαπιστώσετε ότι έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα εκεί. Ε, Έχουμε να χρησιμοποιούμε τη διαδικασία του REFIT ε, για, τη, για διάφορα νομοθετικά κείμενα που έχουν σχέση με, την, το περιβάλλον και θα ήθελα να πω το εξής. Δεν θα πρέπει ε, το ε, κεκτημένο να αμφισβητηθεί. Θα πρέπει να κινηθούμε ακόμα πιο μακριά για τα θέματα της βιοποικιλότητας. Δεδομένης της απειλής και το κινδύνου που αντιμετωπίζουμε. Σας ευχαριστώ για την ε, ενωτική αριστερά Κατερίνα Κονέτσα. Ευχαριστώ. Το είπατε κι εσείς κύριε Αντιπρόεδρε στην αρχή της ε, εισαγωγής σας. Ε, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός θεμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητές σας και μας αφορούν. Η αρχική σας ε, εισαγωγή έκανε λόγο για συνένεση. Όμως, βλέποντας τα πρώτα σας βήματα, τις πρώτες σας αποφάσεις, και βλέποντας επίσης και το πόσο καθυστερήσατε να ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας, τρεις μήνες συγκεκριμένα, αρχίζω να αμφιβάλλω. Βλέπουμε ότι ως τμήμα της διαδικασίας REFIT ε, έχετε αποσύρει νομοθετικά κείμενα χωρίς να ρωτήσετε τη γνώμη μας. Αυτό πιστεύετε ότι είναι καλό σημείο εκκίνησης για τα επόμενα πέντε χρόνια στα οποία θα συνεργαστούμε. Δεν πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο βλάπτει τις ε, σχέσεις μεταξύ μας. Κατά την άποψή μου δεν είναι ορθή πολιτική απόφαση. Αντί να αποσύρεται νομοθεσία θα έπρεπε να εστιάσουμε στην εφαρμογή της νομοθεσίας που ήδη υφίσταται στα κράτη-μέλη. Είναι γνώση μας ένας μεγάλος αριθμός περιπτώσεων που η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν εφαρμόζεται και μάλιστα συχνά εις βάρος της υγείας των πολιτών. Δεν θα ήταν λοιπόν καλύτερα ε, να ε, σιγουρέψουμε την εφαρμογή της νομοθεσίας αντί να αποσύρουμε κείμενα τα οποία θα βοηθούσαν την ε, διατήρηση του περιβάλλοντος. Τώρα, για την ε, TTIP, την ε, Διατλαντική ε, Συμφωνία. έχετε μιλήσει για την ανάγκη του διαλόγου, της σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. Πιστεύετε ότι ως τμήμα του διαλόγου και του δικαιώματο πληροφόρηση θα ήταν καλύτερα οι λαοί μας να γνωρίζουν περισσότερα για την ε, συμφωνία TTIP αντί να τα μαθαίνουν από διαρροές στον τύπο κλπ. Είπατε για, μιλήσατε για διάλογο. Αυτό θα ήταν τμήμα μια τέτοια διαδικασίας. Ενημέρωση των πολιτών. Σας ευχαριστώ. Ε, για τους πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Επιτροπέ που ήρθατε. Χαίρομαι γιατί δεν είχατε έτσι ένα έτοιμο γραπτό λόγο, είστε ανοιχτό στο διάλογο και αυτό είναι πολύ καλό. Γι' αυτό θα ήθελα εγώ να αναφερθώ σε τρία πράγματα που αναφέρατε στην εισαγωγή σας και που νομίζω ότι πρέπει να τα προσέξουμε λίγο. Πρώτα απ' όλα ε, είπατε ότι η καλύτερη νομοθεσία δεν έχει καλό, καλή εικόνα αλλά μάλλον εσείς συμβάλλετε, εσείς ή εγώ λέει ο, πρόεδρο, ο συμβάλλετε σε αυτή την κακή εικόνα. Ναι, ίσως όλοι μας, δεν ξέρω. Ε, ε, ε, στην ουσία συζητήσαμε ας πούμε για το θέμα του ρίφετ αλλά τελικά το ξεχάσαμε δεν επίσης ορίσατε τον Στόιμπεχ ως υπεύθυνο για την καλύτερη νομοθεσία γνωρίζοντας ότι είναι αμφιλεγόμενο άτομο και τελικά οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και οι οργανώσεις των πολιτών, τα συνδικάτα ε, δεν τον ήθελαν και παρόλα αυτά τον ορίσατε τελικά ε, σε μια ακόμα ψηλότερη θέση ως ειδικό σύμβουλο. Γιατί το κάνατε αυτό, εξηγήστε μας. Δεύτερον, μας είπατε ότι σας ενδιαφέρουν πολύ τα αποτελέσματα. Δεν σας ενδιαφέρει μονάχα, ε, μάλλον δεν σας ενδιαφέρουν μόνο οι στόχοι, αλλά και η μεθοδολογία της επίτευξης των στόχων. Καλύτερη νομοθεσία, συχνά διαβάζετε ότι θεωρείτε ότι τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο ε, πρέπει να συμπληρώνουν το ένα το άλλο. Δηλαδή βάζουμε ένα, μια καινούργια, ένα καινούργιο νομοθέτημα και αφαιρούμε ένα. Ε, στην ουσία όμως ε, δεν κάνετε αυτό που ευαγγελίζεστε, δηλαδή στην ουσία αντί να έχουμε έναν ευρωπαϊκό ε, κανόνα αντί για 29 ε, ευρωπαϊκούς, εθνικούς, ε, κάνετε το ανάποδο. ναι, αυτό που μας ενδιαφέρει ε, είναι να δούμε τι συμβαίνει και στις διάφορες χώρες και τι κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτού του είδους ε, η πρόταση μερικές φορές είναι λίγο ανόητη. Επίσης αναφερθήκατε στην συνεκτικότητα και στη συνοχή. Στην, στο έγγραφο για την Ενεργειακή Ένωση γίνεται λόγος ε, για τα απόβλητα της ενέργειας. Αυτή τη στιγμή δηλαδή κάνουμε τώρα κάποιες ε, προτάσεις. Έχει αποσυρθεί η πρόταση για την κλική οικονομία. Είπατε ότι θα υπάρξει αργότερα καλύτερη νομοθεσία. Οκ, εντάξει, το δέχομαι. Αλλά παρόλα αυτά ε, το πιο ηλίθιο πράγμα που μπορεί κανείς να κάνει με τα απόβλητα ε, μετά από το χειρότερο που είναι το να τα θάψει κανείς σε χωματερές είναι ε, να τα κάψει και εσείς βλέπουμε ότι προωθείτε την αποτέφρωση και δίνεται ένα εσφαλμένο μήνυμα λέγοντας προς τις εταιρείες ανακύκλωσης και προς την ανακύκλωση γενικότερα ότι δεν θα υπάρξει πρόθεση της ανακύκλωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την Ευρώπη της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. Ε, θα μιλήσω στα Ιταλικά, πολύ ωραία. Κύριε Επίτροπε, εγώ θα ήθελα να προσθέσω ένα ερώτημα αναφερόμενος σε αυτά τα οποία ήδη αναφέρθηκαν όσον αφορά την, την απόσυρση νομοθετικής πρότασης για τα απόβλητα. Ε, κατάλαβα ότι αυτό αφορά όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος, δηλαδή ότι η Κομισιόν δεν λαμβάνει ε, υπόψη της ως πρωταρχική σημασία στο θέμα των αποβλήτων και δεν θεωρεί καν ότι είναι επίγον το θέμα, αλλά αν αυτό δεν είναι επίγον πέστε μου ποιο είναι πιο επίγον. Εγώ ζω σε μια χώρα όπου όλα, όλοι οι θεσμοί μαζί με την αστυνοπία και, τα και όλοι τέλος πάντων ε, οι φορείς επέτρεψαν φορτηγά να ξεφορτώνουν απόβλητα ε, στην χώρα μου. Επίσης ε, να ρίχνουν σκουπίδια σε καλλιεργήσιμες γέες τις οποίες παραχωρούσαν οι γεωργοί γιατί είχαν οικονομικό πρόβλημα. Πέστε μου, είναι δυνατόν ε, να μην είναι επίγον ένα θέμα το οποίο αφορά εκατομμύρια ευρώ τα οποία, ε, ε, τα, οποία χρησιμοποιήθηκαν, δαπανήθηκαν έτσι ώστε εν τέλει το υλικό οικολογικής ανακύκλωσης απλώς να αποτεφρώνονται και οι τέφρες να ρίχνονται σε ολόκληρες περιοχές, καλλιεργήσιμες γης κλπ η ίδια η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας μαζί με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν ε, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι καρκινογένειες, διάφορες ασθένειες, ε, ε, σχηματισμοί και παραμορφώσεις εμβρίων οφείλονται σε αυτήν την κακή διαχείριση των αποβλήτων. Δεν είναι επίγον αυτό. Ευχαριστώ πολύ θα δώσω αμέσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο ε, Τίμερμαν, έτσι ώστε να δώσει μία πρώτη απάντηση σε αυτό το πρώτο γύρο των ερωτήσεων. Ευχαριστώ. Why did we meet? Ευχαριστώ. Καταρχήν γιατί η συνάντηση γίνεται τώρα. Καταρχήν κύριε Λίζε, ε, είσαι από τους πρώτους με τους οποίους συναντήθηκα. Και πάνω από μία ώρα, πάνω από μία μισή ώρα νομίζω συζητήσαμε όλα αυτά τα θέματα. όχι μόνο με εσάς και με αρκετούς συναδέλφους σας συναντήθηκα. Πάντως, σοβαρά τώρα, ήθελα να γίνει αυτή η συνάντηση με την Επιτροπή σας. Και νομίζω σχεδόν κανένας άλλος Επίτροπος δεν έχει συναντήσει τόσε πολλέ επιτροπέ όσε εγώ ή τόσους πολλούς Ευρωβουλευτές όσους εγώ. Είναι πολλές Επιτροπές, επιτροπέ, κάνω ό,τι μπορώ και χαίρομαι ιδιαίτερα που μα δίνει τη ευκαιρία να συναντηθούμε έστω και τώρα. Ελπίζω να το αποδέχεστε ως εξήγηση. Δεν υπήρχε κανένας πολιτικός λόγος να περιμένουμε μέχρι σήμερα. Από τότε που ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής ε, ήταν τόσο έντονες οι εργασίες μας που τουλάχιστον εγώ ήθελα πάρα πολύ να συναντηθώ με την Επιτροπή σας το συντομότερο δυνατόν. Δεν υπήρχε κανένα πολιτικό ζήτημα που εμπόδισε το να γίνει η, Επιτροπή, η συνάντηση αυτή νωρίτερα, κάθε άλλο. Όπως αναφέρατε και εσείς στην παρέμβασή σας, υπάρχουν πολλά τα θέματα στα οποία θα ήθελα να κάνουμε ανταλλαγή απόψεων. Για το πακέτο τώρα για τα απόβλητα υπάρχουν ε, πολλά ε, στοιχεία και θα ήθελα να το συζητήσουμε. Καταρχήν, πιστεύω ότι αν ε, προσπαθήσουμε και δουλέψουμε σκληρά, θα μπορέσουμε να υποβάλουμε ένα πλήρες πακέτο για την κυκλική οικονομία και συγκεκριμένα για τα απόβλητα θα υποβάλουμε μία αναθεωρημένη πρόταση κατά τρόπον ώστε τελικά να μην έχει χαθεί καθόλου χρόνος από τη στιγμή που είχε υποβληθεί αρχικά αυτό το πακέτο μέτρων. Ο κ. Σέκχαουτ ανέφερε αρκετούς λόγους και για όλους αυτούς τους λόγους ε, καλό είναι να επανεξεταστούν οι προτάσεις ο κίνδυνος ε, του να καταφύγουμε στην ε, ε, κάθεση των απορριμμάτων στην τωρινή δέσμη μέτρων ήταν ένας κίνδυνος που έπρεπε να λάβουμε σοβαρά υπόψη μα. Μας είπαν ότι αν το κάνετε έτσι, διατρέχετε τον κίνδυνο. ακριβώς όπως το περιέγραψε ο κύριο Άικχαουτ αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε, δηλαδή το να οθήσουμε ορισμένα κράτη-μέλη στο να αυξήσουν το δυναμικό αποτέφρωσης απορριμμάτων αντί να αναζητήσουν πιο βιώσιμες λύσεις. Ήταν λοιπόν ένας από τους λόγους για τους οποίους έπρεπε να αναθεωρηθεί αυτή η δέσμη μέτρων. Καταρχήν λοιπόν η ποιότητα της νομοθεσίας ήταν αυτό που έπρεπε να φροντίσουμε. Δεύτερον, κάτι το οποίο έχω ήδη συζητήσει με πολλούς ε, ενδιαφερομένους για το θέμα αυτό και στον Ταβός, το αναφέρατε και εσείς στον Ταβός, είπα συγκεκριμένα ότι αν θέλετε να έχετε μία ε, συνεπή πρόταση για την κυκλική οικονομία θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλοι οι τομείς, όχι μόνο τα απορρίμματα. Και ένας από τους ε, συγγραφείς του βιβλίου Cradle to Cradle προσφέρθηκε να δουλέψει μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τα χαράς δεχτήκαμε την προσφορά του. Και ο συνάδελφος Επίτροπος Μέντες ε, ζήτησε από τη βιομηχανία να μας ε, υποβάλει προτάσεις για το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε μια κυκλική οικονομία πλήρη. και να μην χρησιμοποιούμε ε, στον κύκλο της παραγωγής μη βιώσιμα προϊόντα, ούτω ώστε να έχουμε μια, έναν πλήρη κύκλο και να μην παράγονται καθόλου απόβλητα από την όλη διαδικασία. Και ότι ο Πρόεδρος Κατάινεν και εγώ και όλοι οι αρμόδιοι επίτροποι καταβάλουμε κάθε προσπάθεια και συνεργαζόμαστε για να έχουμε τελικά μέσα στο 2015 ένα πλάνο. Θέλουμε να το κάνουμε μέσα στην τωρινή χρονιά και να μην χάσουμε καθόλου χρόνο. Δεν θέλω λοιπόν να υπάρχει κανένα σημείο παρανόησης. Είναι πολύ επίγοντα να κάνουμε κάτι για τα απόβλητα. Το γνωρίζει η Επιτροπή ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με τρόπο βιώσιμο. Και αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν προβληματικές λύσεις για το περιβάλλον ε, εξίσου προβληματικές με τις ε, χωματερές. Ε, δεύτερο θέμα, οικολογικός σχεδιασμός. Επανεξετάζουμε τη δέσμη μέτρων για τον οικολογικό σχεδιασμό, όχι αλλάζοντας τους στόχους, οι στόχοι θα παραμείνουν. και με τον κύριο Λίζε το είχαμε συζητήσει όταν πρώτο συναντηθήκαμε. Πρέπει να δούμε αν το προτινόμενο μέτρο είναι το βέλτιστο μέτρο που θα μας οδηγήσει εκεί που θέλουμε. Ο οικολογικός σχεδιασμός πολλές φορές έχει οδηγήσει στην εξοικονόμηση ενέργειας και ακριβώς αυτό επιθυμούμε. Θα είμαστε λοιπόν πολύ προσεκτικοί στο πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Ε, χαίρομαι που ο κύριος Κρότε είπε ότι πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον. Ακριβώς αυτό θέλουμε να εξετάσουμε με την κυκλική οικονομία ε, και τη δεσμή σχετικά με τα απορρίμματα. Και όταν μιλάμε με διευθύνοντες συμβούλους μεγάλων ε, εταιριών, αυτό λέμε. και με τους ακαδημαϊκούς αλλά και με τους κύκλους ε, της βιομηχανίας ε, όλοι συμφωνούμε ότι είναι ιδιαίτερα ε, ενδιαφέρουσα η κυκλική οικονομία καθώς και αναπόφευκτη. Και εκεί γίνεται, αναγνωρίζεται περισσότερο αυτό το θέμα παρά μεταξύ των πολιτικών. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι από όλους τους τομείς της οικονομίας να συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια όλοι όσοι πιστεύουν ε, στα ωφέλη που έχουμε από την κυκλική οικονομία και με τη βοήθειά τους ε, να συνεργαστούμε και να γίνουμε πραγματικά ηγέτες ε, στην παγκόσμια αγορά σε αυτά τα θέματα. Χώρες όπως η Κίνα, ακόμη και η Κίνα, αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνονται τα ωφέλη της κυκλικής οικονομίας και εμείς μπορούμε να είμαστε παγκοσμίω πρώτοι που θα το ε, θέσουμε και θα το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και με το πρόγραμμα Juncker θα μπορέσουμε να επενδύσουμε στην κυκλική οικονομία και μέσα στους επόμενους μήνες ελπίζω να έχουμε αυτή τη δέσμη μέτρων για να σας δείξουμε και τα πρώτα αποτελέσματα. Ένα σημαντικό θέμα είναι και το ότι σε εθνικό επίπεδο δεν γίνεται η μεταφορά της νομοθεσίας πάντοτε κατά το βέλτιστο τρόπο και πολλές φορές ε, ότι έχουμε υπερθεματισμό κανονιστικών διατάξεων. Προσπαθούμε πολλές φορές να αντιμετωπίσουμε την κρίση και δεν ελέγχουμε την τελική εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνουμε. Πρέπει να είναι σαφές ότι η Επιτροπή είναι υπέρ ε, της σωστής εφαρμογής, γιατί αν ε, οι φορείς της αγοράς πιστέψουν ότι η Επιτροπή δεν θα ασχοληθεί με τη σωστή υλοποίηση των μέτρων που προτείνουμε, αυτό θα είναι εις βάρος όχι μόνο του περιβάλλοντος, αλλά θα χάσουμε και πολλές οικονομικές δυνατότητες και ευκαιρίες. Μας ανησυχεί λοιπόν αυτό το θέμα της σωστής ε, μεταφοράς κοινοτικού δικαίου σε εθνικό δίκαιο και κάθε φορά που έχω επαφές ε, στα κράτη-μέλη με επιχειρήσεις, με τους οικονομικούς φορείς βλέπω ότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ ο τρόπος με τον οποίο ε, υλοποιούνται στην πράξη τα μέτρα τα οποία εμείς θεσπίζουμε. Υπάρχει τεράστια απόσταση μεταξύ ημών σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα κράτη-μέλη. Είναι μεγαλύτερη αυτή η απόσταση από ό,τι μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και της ευρωπαϊκής ε, βιομηχανίας. Αυτό το οποίο θα θέλαμε είναι το να κλείσουμε, ε, να μειώσουμε αυτή την απόσταση μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν υπάρχει καμία επιθυμία να αντιβούν προς τις διατάξεις σχετικά με την αηφόρο ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα. Κάθε άλλο. Θα δείτε ότι σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη-μέλη και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ξεκινούν πολλά τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας ενδιαφέρει λοιπόν πάρα πολύ το να έχουμε την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και είναι ένας κίνδυνος το να βλέπουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεωρούν την Ευρώπη κάτι το δίσκαμπτό και δύσκολο να υλοποιηθεί και μερικές φορές ε, ε, απομακρύνονται από τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί ακριβώς μας θεωρούν κάτι απομακρυσμένο και αυτό είναι μια τάση που πρέπει να ε, αντιστρέψουμε. Μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι ε, ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε όταν θέλουμε να θεσπιστεί κάτι στις οδηγίες μας. Θέλουμε να υπάρχει σαφήνεια για το στόχο που θέλουμε να επιτύχουμε και αφήνουμε στα κράτη-μέλη τη διακριτική ευχέρεια να αναζητήσουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να υλοποιήσουν αυτά τα οποία εμείς θεσπίζουμε. Πολλές φορές όμως με το πέρασμα του χρόνου διαπιστώνουμε ότι οι ίδιες οι οδηγίες ε, γίνονται πολύ ρυθμιστικές, υπερβολικά ρυθμιστικές θα έλεγα, για το πώς θα υλοποιήσουν συγκεκριμένα τα κράτη-μέλη αυτές τις διατάξεις. Και εδώ πάλι θα πρέπει τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ο διοργανικός διάλογος να βοηθήσει την καλή νομοθεσία και να διευκρινίσουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε σωστά τα νομοθετικά μέτρα που έχουμε στη διάθεσή μας βάσει των συνθήκων. Σε πολλούς τομείς θα πρέπει να τονίζουμε τους στόχους μας και να μην είμαστε υπερβολικά ρυθμιστικοί εξηγώντα τα κράτη-μέλη πώς ακριβώς θα υλοποιήσουν αυτούς τους στόχους. Και αυτό είναι κομμάτι αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε με την ε, καλύτερη νομοθεσία. Και για την Ενεργειακή Ένωση συγκεκριμένα, για να μπορέσει να είναι επιτυχημένη, δεν μπορεί να πρόκειται μόνο για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και των προμηθευτών. Θα πρέπει να ε, μας απασχολήσει η μετάβαση. Θα πρέπει ε, οπωσδήποτε να μιλήσουμε για τη μεταβατική, ε, για τη φάση της μετάβασης σε άλλες ενέργειες πέραν των ορεικτών καθήμων. Και χρειάζεται μια συνεκτική προσέγγιση σε όλους τους τομείς. Νομίζω ότι αν θελήσουμε να γράψουμε ένα έγγραφο για την βιώσιμη ανάπτυξη και μόνο δεν σημαίνει ότι ενοποιούμε τις προσπάθειές μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ε, θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και πάλι σαν ε, μια απομονωμένη προσπάθεια. Ενώ εμείς θέλουμε η προσπάθεια αυτή να ενταχθεί σε όλες τις άλλες προσπάθειες ε, νομοθεσίας. Αφήσαμε λοιπόν να το συζητήσουμε με τους συναδέλφους μου για να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή λύση. Για την βιοπικιλότητα θα επανέλθω, δεν είμαι ενημερωμένο, δεν θέλω να σας δώσω ε, μια ουδέτερη απάντηση, θα σας απαντήσω γραπτός. Σε ό,τι αφορά την διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι διαβουλεύτηκα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζήτησα τη γνώμη σα και η γνώμη σα ήταν πολύ σαφή και με διάφορου τρόπου. Εκφράσατε την άποψή σα για το πρόγραμμα εργασία τη Κομισιόν. Ο κ. Λίζα μάλιστα ήταν πολύ ειλικρινή. Ε, ο ίδιος έχει μια άποψη, αλλά ενδεχομένως η πολιτική του ομάδα έχει μια άλλη. Και εγώ πρέπει να λάβω υπόψη τη γνώμη της πλειοψηφίας. Υπέβαλα το πρόγραμμα ε, δράσης κομισιών, άκουσα την, τις απαντήσεις, αλλά ε, δεν είχαμε κάποια συγκεκριμένη πλειοψηφία. Εγώ άκουσα την γνώμη του Κοινοβουλίου και στην Ολομέλεια και αλλού και στις πολιτικές ομάδες, γιατί επισκέφτηκα όλες τις πολιτικές ομάδες. Οπότε δεν είναι σωστό να λέγεται ότι δεν διαβουλεύτηκα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την TTIP, την Διατλαντική Εμπορική Συμφωνία. Είμαστε πάρα πολύ διαφανείς, πιο διαφανείς από οτιδήποτε άλλοτε στο παρελθόν. Μία από τις πρώτες αποφάσεις της Κομισιόν, αυτή της Κομισιόν, ήταν μεγαλύτερη διαφάνεια στα έγγραφα ε, τα οποία συζητούνται κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Οπότε δεν καταλαβαίνω αυτό που λέγεται ότι ε, οι πολίτες ενημερώνονται και εσείς ενημερώνεστε μόνο μέσω διαρών. Κύριε Στόιμπερ, ο κ. Στόιμπερ είναι ε, σύμβουλος των πρόεδρων της Κομισιόν. Κάθε μέλος της ε, Κομισιόν, κάθε επίτροπος έχει το δικαίωμα να διορίσει ένα αριθμό συμβούλων. Ο κ. Στόιμπερ είναι ένας από τους συμβούλους του Προέδρου, όπως και ο κ. Μπαρνιέ για παράδειγμα. Και εγώ έχω ένα αριθμό συμβούλων και ο κ. Στόιμπερ ο κ. Στόιμπερ θα ε, μοιραστεί μαζί μας ε, την μακρόχρονη εμπειρία του. Είπα όμως και έχω πει και το επαναλαμβάνω ε, όταν προγραμματίζω την βελτίωση της νομοθεσίας θα ε, φροντίσω, θα μεριμνήσω έτσι ώστε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να ε, πούν τη γνώμη τους. Θα ακούσω και τις βέλτιστες πρακτικές, τις καλύτερες εμπειρίες στα κράτη-μέλη. Ε, άλλοι λένε ότι το ένα παραπάνω, ένα λιγότερο είναι το καλύτερο. Ε, άλλοι λένε ότι σε οτιδήποτε επιτυχάνει σε, ευρωπαϊκό, σε εθνικό επίπεδο δεν λειτουργεί απαραίτητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακούω πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, ε, θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι η Εθνική Νομοθεσία θα έχει ρήτρε ε, ολοκλήρωσης, ρήτρε κατάργησης, έτσι αυτό θα επέβαλε στις εθνικές κυβερνήσεις να ξαναδούν την ομοθεσία αυτή κάποια στιγμή στο μέλλον, πράγμα το οποίο δεν κάνουν πολύ συχνά. Νομίζω ότι απάντησα στις ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις λεπτομερείς απαντήσεις. Τώρα αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα. Έχω 26 αγορητές εγγεγραμμένους, ο αντιπρόεδρος θα πρέπει να φύγει στις 8 και 20. Επομένως θα ήθελα να σας παρακαλέσω κάθε ερώτησή σας να είναι ε, ένα λεπτό. Θα ξεκινήσω αμέσως με τον Ιβο Μπέλετ. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, θα μιλήσω Ολλανδικά και είναι πιο απλό για να κατανοήσουμε ο ένας τον άλλον. Αναφερθήκατε στην κυκλική οικονομία, και εγώ θέλω να κάνω ακόμα μια ερώτηση για να συμπληρώσουμε το θέμα. Όταν αναφέρεστε σε αυτή την πολιτική ανακύκλωση, άλλωστε είπατε και στην ακρόαση ότι δεν πρόκειται για απόβλητα ε, αλλά για αξιολόγηση ε, των ε, μάλλον αλλά πρόκειται για μια διαδικασία που θα δώσει αξία και στα απόβλητα και θα δημιουργήσει κάποια νέα υλικά. Ε, και πρόκειται για υλικά τα οποία ενδεχομένως θα εξαχθούν ε, ε, και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό, γιατί δεν τα κρατάμε εμείς, δεν έχουν τόσο μεγάλη αξία. Δεύτερον, προστασία καταναλωτού. Είναι και αυτό στο ευρύ χαρτοφυλάκιό σας. Αληθεύει ότι ε, ε, προτίθεστε να κάνετε κάποιες, να αναλάβετε κάποια μέτρα όσον αφορά κυρίως την προστασία των νέων, την προστασία της υγείας των νέων. Ε, νομίζω ότι ε, περιμένουμε κάποιο νομοθέτημα όσον αφορά την προστασία των νέων επίσης ε, στα πλαίσια της ψηφιακής κοινωνίας. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω όσον αφορά τα θέματα αυτά. Να μην ξεπερνάτε το χρόνο ομιλία σας παρακαλώ. Um, Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Είπατε προσφάτως σε μια συνομιλία με τον Ρόδο ότι δεν ήταν ιδεολογική η προσέγγιση σας για την μείωση της γραφειοκρατίας. Και αναφέρετε και τώρα ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις φοβούνται τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται η νομοθεσία. Κάτι που μας ανησυχεί είναι ότι μέχρι τώρα είχαμε έναν τρόπο λειτουργίας ε, η φετινή χρονιά είναι κέρια σημασία ε, για την κλιματική αλλαγή. Υπάρχει δέσκεψη στο Παρίσι και για την ανάπτυξη έχουμε το Σεπτέμβριο της ε, συναντήσεις και αφορούν και εμάς και την Επιτροπή Ανάπτυξης. Τι διασφαλίσεις μπορείτε να μας δώσετε για να απαλύνετε τους φόβους σας, τους φόβους μας. Πώς μπορείτε να μας καθησυχάσετε ότι όντως αναλαμβάνετε μια δέσμευση να έχουμε νομοθεσία που θα ε, διασώσει τις βασικές περιβαλλοντικές προτεραιότητες ε, που ήδη υπάρχουν. Ευχαριστώ. Κύριε Σνέκερ, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε, χαίρομαι που είστε σήμερα κοντά μας. Εξαιρετική ευκαιρία να έχουμε ανταλλαγή απόψεων και να μιλήσουμε για την κυκλική οικονομία. Ως σκιώδης ηγητής από το ECR έχω μια συμπληρωματική ερώτηση. Την περασμένη Τετάρτη κάναμε μια συζήτηση σε, σε, σχέση και με την Φλάνδρα που είναι η περιοχή την οποία και εγώ εκπροσωπώ. Επισκεφτήκαμε ε, κάποιες εγκαταστάσεις που αποτελούν και βέλτιστες πρακτικές και έχω και συγκεκριμένες ερωτήσεις που προέκυψαν. Συμφώνησαν όλοι ότι η εσωτερική αγορά ήταν απολύτως απαραίτητη και ότι οι ευρωπαϊκοί μας στόχοι θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τους στόχους της εσωτερικής αγοράς. Δεν υπάρχουν όμως οι προϋποθέσεις ε, για δίκαιο ανταγωνισμό ακόμη. Θα έπρεπε η Επιτροπή μερικές φορές να είναι πιο συγκεκριμένη ανακράτως μέλος. Πώς θα μπορούσατε να το κάνετε και πώς θα μπορούσατε να συνεισφέρετε στη δημιουργία ενός ε, πεδίου δίκαιου ανταγωνισμού. Μια δεύτερη ερώτηση για την κυκλική οικονομία. Σαφώς χρειάζεται ανταγωνιστική αγορά και εταιρείε που θα λειτουργούν μέσα σε αυτή την ανταγωνιστική αγορά. Πώς θα προωθήσετε την ανακύκλωση στην πραγματικότητα. Και μια ακόμη ερώτηση σε σχέση με αυτό που είπε και ο Ήβο προηγουμένως. Ήδη υπάρχει σπάνης πρωτογενών προϊόντων και δεν έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλά προϊόντα τα οποία πρέπει να εισάγουμε. Δεν έχουμε λοιπόν στρατηγικά από θέματα στρατηγικές προμήθειες που χρειάζονται οι βιομηχανίες μας. Αυτό πώς θα το αντιμετωπίσετε. Κυρία Μπέρντερ, ένα λεπτό. Κυρία Μπέρντερ, ένα λεπτό. Πέρσι στηρίξαμε με μεγάλη πλειοψηφία το αίτημα να υποβάλλεται πρόγραμμα δράσης για, τα, ε, για την καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά των, της Άγριας Πανίδας που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, ένα εμπόριο πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια ε, το χρόνο. Ε, είναι ένα πρόβλημα το οποίο ε, καταλαβαίνω και ψηλότερη στην διεθνή ατζέντα. Ε, τόσο στην Κίνα όσο και στις νομές Πολιτείες επιβάλλονται περιορισμοί στις ε, εισαγωγές είδων προκύπτων από αυτό το, ε, το, τα εγκλήματα κατά της Πανίδας. Ε, πιστεύω ότι εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, περιθώριο να δράσει. Ως αντιπρόεδρος θα στηρίζατε την, τον Επιτροπό αν ε, υπέβαλε προτάσει για αυτό το θέμα. Είναι ένα ζήτημα για το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δράσει εδώ και τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι αντικαταστάτρια ε, από την Επιτροπή Ίντα ε, και με ενδιαφέρουν τα ζητήματα διεθνούς εμπορίου. Θα ήθελα να θέσω τις ίδιες ερωτήσεις που έθεσαν και κάποιοι προηγούμενοι συνάδελφοι. Η περίπτωση Vattenfall ε, εναντίον Γερμανίας, για παράδειγμα, ε, πρόκειται για θέμα απαγόρευση χρήση συγκεκριμένων τύπων ενέργειας δεν πιστεύω ότι οι κάτω θα πρέπει να πάρουν παρόμοια απόφαση. Ο Γιούνκερ ε, είπε ότι δεν θα πρέπει να υπογραφεί η συμφωνία TTIP αν δεν συμφωνεί η Γαλλία. Θα κάνετε κάτι για αυτό το θέμα. Thank you very much. And now Η βελτίωση της ε, νομοθεσίας ε, δεν σημαίνει απλώς ε, καλύτερα έγγραφα, αλλά και καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας. Οι εγγυήσει εφαρμογής είναι τμήμα του συστήματος ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που, η οποία ελέγχει την σωστή μεταγραφή Χρειάζεται όμως ε, τα κράτη-μέλη να διαθέτουν και ισχυρούς θεσμού και βέβαια η Κομισιόν να είναι σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη προκειμένου να ελέγχεται η σωστή μεταγραφή και εφαρμογή της νομοθεσίας. Ο κ. Ποτότσνικ, ο προηγούμενος Επίτροπος Περιβάλλοντος, είχε ξεκινήσει κάποιες πρωτοβουλίες για ε, ε, τη χρήση τη δικαιοσύνη και της επιθεωρη, περιβαλλοντικής Η Κομισιόν τώρα τι θα κάνει σε ό,τι αφορά τις ε, περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις και την πρόσβαση στην ε, δικαιοσύνη. Ε, Σας ευχαριστώ, η συνάδελφος Εύη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ, όπως και άλλοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ στα πρόσφατα δημοσιευθέντα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, όπου αναφέρεται ότι 14 δείκτες που λαμβάνονται υπόψη και ε, βράχη και μέσο και μακροπρόθεσμα ε, οι τροποποιήσεις ε, είναι πάρα πολύ αρνητικές. Μεταξύ των δικτών σε επιδείνωση, ε, είναι διάφορα, ε, διάφορες ε, παράμετροι που αφορούν ας πούμε την βιοπικιλότητα, την, ε, τα αέρια του θερμοκηπίου, ε, πανίδα χλωρίδα κτλ. Επίσης, εκτός από ε, την ε, τους δείκτες αυτούς ε, έχουμε και μία σειρά μελετών που δείχνουν ότι πάνω από 400 ασθένειες, ε, συγγνώμη, πάνω από 400 είναι οι θάνατοι οι οποίοι άμεσα σχετίζονται με τους διαταράκτες, ορμονικούς διαταράκτες, χημικές ουσίες οι οποίες τροποποιούν το ορμονικό σύστημα κτλ. Ε, δεν ε, έχουμε ένα σχετικό έγγραφο από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος ε, που μας είχατε υποσχέσει ότι θα το έχουμε και τελικά δεν το έχουμε στη διάθεσή μας. Μπορείτε να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Ο κύριος Φλόενς. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Χαίρομαι που είστε κοντά μας και καλωσορίσατε. Δεν θα διαφωνήσουμε, έχουμε διαφωνήσει αρκετά στο παρελθόν. Άκουσα ε, αυτά τα οποία είπατε για την πολιτική, συγκεκριμένα ε, βήματα τα οποία θα αποτελέσουν την πολιτική σας. Μου άρεσε και το παράδειγμα που δώσατε με τα σιλό που είπατε ότι κάθε πολιτική από κάθε μέτρο αποτελεί ένα σιλό, ένα μεμονωμένο τομέα ενώ θέλετε η βιώσιμη ανάπτυξη να είναι κάτι που διέπει όλους τους ε, τομείς. Όμως πώς θα φτάσετε στο αποτέλεσμα της ε, καλής νομοθεσίας. Θα θέσετε δεσμευτικούς στόχους και συνάδελφοι από το ECR ε, το ανέφεραν. Υπάρχουν ε, πολλοί στόχοι τους οποίους θέτουν διάφορες κυβερνήσεις και η δική μας στη χώρα μας. Πώς όμως μπορεί η Επιτροπή να συγκρίνει τους συγκεκριμένους στόχους που θέτει κάθε χώρα. Θα μπορέσουμε ίσως να τα συζητήσουμε ίσως ε, και με ένα ποτήρι μπύρα. Ευχαριστώ. Αντιπρόεδρος Πανιό. Κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, άκουσα ένα μέρος της ε, παρέμβασή σας με μεγάλη χαρά. Και με την ίδια χαρά θα ήθελα να σας υποβάλω ένα ερώτημα. Πολύ σύντομο. Εδώ και λίγο καιρό προωθείται ε, η τροποποίηση της ε, διαφάνειας ε, του καταλόγου των ομάδων πίεσης των λόμπι που είναι παρόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρώτος κανόνας λοιπόν λέει ότι πρέπει να, καταγράφονται αυτά τα λόμπι. Έχουν καταγραφεί ήδη 966 τέτοια λόμπι Εσείς θέλετε να προχωρήσετε από ό,τι φαίνεται. Ε, και ε, να παρουσιάσετε τη συμφωνία αυτή ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αληθεύει αυτό και πότε θα το κάνετε γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε ένα ακόμα βηματάκι στην πολιτική διαφάνεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η κυρία Σερή Πιερίτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερος ευτυχής που συναντώ τον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς εδώ. Άκουσα με μεγάλη προσοχή ε, ε, τα όσα αναφέρθηκαν για την οδηγία ε, Habitat. Βλέπω τις κάτω χώρες ας πούμε και την υλοποίηση της οδηγίας Habitat σε διάφορους τομείς βλέπω ότι ε, υπάρχουν ε, πολλοί περιορισμοί, αλλά στο άρθρο 2, παράγραφος 3, αναφέρεται, ε, γίνεται αναφορά στις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένη ερώτηση λοιπόν και φαντάζομαι ότι την περιμένατε τι γίνεται τώρα στην ε, Ευρώπη. Ε, γίνεται μία προσπάθεια ε, να τροποποιηθεί η οδηγία Habitat, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουν κάποια σημαντικά σημεία της πώς θα κινηθείτε έτσι ώστε όσο γίνεται πιο γρήγορα να γίνει ένας κατάλογος. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Μποναφέ. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτά που μας είπατε ε, νομίζω ότι ήταν ε, μουσική στα αυτιά, τα δικά μου και ε, άλλων. Γιατί μας είπατε ότι η βιωσιμότητα θα αποτελέσει το κεντρικό άξονα πάνω στον οποίο θα βασιστούν και άλλες πολιτικές. Νομίζω ότι όλοι θέλουμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη της οικονομίας μας. Είναι σημαντικό πάντως ότι το παλιό μοντέλο ανάπτυξης ε, δεν λειτουργήσε καλά και επομένως ε, είναι σαφές ότι ε, στο κέντρο των νέων πολιτικών θα πρέπει να βρίσκεται ακριβώς αυτή η λέξη, η βιωσιμότητα. Ε, δεν θα πρέπει δε να παρουσιάζεται ως ε, δέσμευση αλλά σαν μια ευκαιρία ε, όπως γνωρίζετε και είδατε και σήμερα για την, για την κυκλική οικονομία είναι γεγονός ότι εμείς έχουμε κάνει πολλή συζήτηση και ξέρουμε ότι μπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη 1% του ΑΕΠ και δημιουργία ενός εκατομμυρίου θέσεων εργασίας. Εσείς μπορείτε σήμερα να μας διασφαλίσετε ότι θα, γίνει, θα γίνουν σεβαστά τα χρονικά περιθώρια και ότι θα υπάρχει πρόταση μέχρι το τέλος του έτους. Επίσης θα είστε πιο ε, φιλόδοξος όσον αφορά ε, την έρευνα ε, η οποία θα είναι συνολική από την αρχή μέχρι το τέλος και από το λίκνο μέχρι ε, το, τον τάφο πιστεύουμε ότι είχαμε φτάσει σε κάποιους καλούς στόχους με την παλιά πρόταση ε, αλλά ε, στην, ε, στη γλώσσα μου λέμε ότι άμα δεν έχεις μπικικίνια τίποτα δεν γίνεται και επομένως εσείς μπορείτε να μας διασφαλίσετε ότι θα δώσετε πραγματικά τη μάχη για αυτήν την αηφόρο βιώσιμη οικονομία. Ευχαριστώ κύριο ε, έχω μια ερώτηση σε 9 τμήματα, θα τολμούσα να πω, αλλά ε, δεν θα ήταν πολύ ευγενικό. Ε, σε ό,τι αφορά την οδηγία τη, για τις μεσέ εγκαταστάσεις ε, καύσης, τι γίνεται με τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ιδιαίτερα σε πλατφόρμες, υπεράκτιες πλατφόρμες, η οδηγία δεν προβλέπει και παρόλα αυτά εφαρμόζονται, εφαρμόζεται αυτή η ε, ε, υποχρέωση περιβαλλοντικών, ε, περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα έπρεπε να αποφεύγουμε τέτοιου είδους εκπλήξεις. Θα Νομίζω θα ήταν λογικό να αφαιρεθούν αυτέ οι εγκαταστάσει από την οδηγία. Θα το υποστήριζα. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να αποφεύγουμε να εκπλήσουμε του ε, συναλλασσόμενου. Ευχαριστώ και Σφαρία. Ευχαριστώ ε, πρόεδρε. Καλώ ήρθατε. Ε, Μα τιμάτε με την παρουσία σα για πρώτη φορά. ελπίζω να ξανάρθετε. Στην προηγούμενη θητεία στήσαμε τη θέση μας για την οδηγία σε ό,τι αφορά την διαφάνεια της τιμής των φαρμάκων. Ως ε, εισηγητής ε, ε, εξασφάλισα μαζί με τους συναδέλφους μου μια μεγάλη πλειοψηφία συναδέλφων. Όμως δεν έχω δει καμία ανταπόκριση από την Κομισιόν. Η Κομισιόν μάλιστα αποφάσισε να αποσύρει την πρότασή της μετά από αντιδράσεις των κρατών μελών. Τα επιχειρήματα της Κομισιόν αρχικά ήταν ότι θα πρέπει να γνωρίζουμε τις τιμές για να καθορίζουμε την συμμετοχή των πολιτών στην αγορά. Ε, ε, θα, επιτρεπώ, θα βοηθούσαμε να, ε, τους ασθενείς να διαθέτουν πιο ε, σύγχρονες με θεραπευτικές μεθόδους και η, θα εξηγέναμε τον τομέα του φαρμάκου. Ρωτήσουμε εξή. Αν αυτά τα επιχειρήματα διατηρούνται, η Κομισιόν έχει σκοπό να ξαναυποβάλει την πρότασή της ε, τροποποιημένη. Και πότε θα γίνει αυτό, Δε, τελευταίο, τέλος. Ποιες θα είναι οι πρωτοβουλίες της Κομισιόν για το πρόβλημα της ε, πρόσβασης σε νέα φάρμακα, για παράδειγμα αυτά της υπατήτητος γάμα. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε παρόσο. Μικρόφωνο παρακαλώ. Μικρό. Perdón, gracias. Ahora. Eh, eh, Κύριε Τίμερμανς, ε, επιθυμείτε να δεν βλέπετε τα πράγματα ολιστικά, με διαβούλευση, ε, πολύ καλό αυτό ως προθέσεις. Ε, δυστυχώς όμως έχω ξεκολουθώ να έχω την εντύπωση ότι ε, πάντοτε περνάτε σε εμά το μπαλάκι. Ε, σαν να μην θέλετε εσείς να είστε αυτοί που θα ξεκινήσουν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες είχαμε, περιμένουμε, ε, λέτε ότι ε, περιμένουμε πρέπει να περιμένουμε όλο το πακέτο για την κοινωνική οικονομία. Όμως αυτό είναι ένα μήνυμα επικίνδυνο που στέλνουμε στους πολίτες. Γιατί τι γίνεται, όσοι ε, επιθυμούν την πρόθεση της ε, καύσης, ε, το, θα έχουν το περιθώριο να το κάνουν. Μετά, σε ό,τι αφορά το δευτερογενές δίκαιο και το ρόλο των κρατών μελών, εσείς επανειλημμένως έχετε πει ότι έχετε μιλήσει με την βιομηχανία να σας ρωτήσω πώς θα λάβετε υπόψη και τη γνώμη των πολιτών καθώς επίσης και των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Ευχαριστώ. Ο κύριος <laughs> ε, ε, Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, αυτή η Επιτροπή έχει θέσει ως βασικές προτεραιότητες τις ε, θέσεις απασχόλησης και την ανάπτυξη. Παράλληλα και με τη βιώσιμη ανάπτυξη, όπως μας είπατε σήμερα. Πώς εξηγείτε λοιπόν τις, ε, την έλλειψη συνέπειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ε, παραμένουν ε, επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα. Θα ήθελα να μας απαντήσετε σε αυτό και σε σχέση με την οδηγία για τα ενδιατήματα των πτηνών. Ε, ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Σουίτσα. Ε, έχω μελετήσει προσεκτικά το, το, συγγνώμη, το χαρτοφυλάκιό σας ε, και ξέρω ότι είστε υπεύθυνο για πολλά πράγματα. Όταν λέτε ότι σε μερικές χώρες οι νόμοι είναι πιο σκληρή ενώ σε άλλες χώρες η προσέγγιση η νομοθετική είναι πιο ήπια ε, δημιουργείται μια αίσθηση ανισότητα στην Ευρώπη. Ε, αλλά πώς ε, μπορείτε κατά την άποψή σας, πώς θα, πώς θα μπορούσαμε να έχουμε πιο συνεκτική προσέγγιση, πώς μπορούμε να φτάσουμε λοιπόν σε μια επιθυμητή συνοχή, λαμβάνοντας πάντως υπόψη ότι κάποιες χώρες μπορούν να συνεχίσουν να νομοθετούν πιο αυστηρά εάν θέλουν. Ε, χαίρομαι επίσης γιατί θεωρείτε ότι η βιωσιμότητα είναι κάτι που αφορά όλες τις ε, πολιτικές. Ο Γιολάινεν. Κύριε Πρόεδρε, Πάντοτε ε, θέλετε ε, τα προγράμματα της Επιτροπής να έχουν πραγματικό περιεχόμενο και έχετε την ευθύνη να το υλοποιήσετε και στα θέματα που αφορούν εμάς. Αποφασίστηκε το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο και η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν για 12 προτεραιότητες ε, μέχρι το 2020. Όλες τις προτεραιότητες θα τις υλοποιήσετε και αν όχι ποιες θα παραλείψετε. Έχουμε συζητήσει πάρα πολύ για την αποδοτικότητα των πόρων, όχι μόνο για την ενέργεια, αλλά και ευρύτερα για την αποδοτικότητα των πόρων και είχε προβλεφθεί ότι θα τεθούν και δεσμευτικοί στόχοι για τη χρήση των υλικών, για τη χρήση της γης και η ερώτησή μου είναι αν όντως πρέπει να περιμένουμε κάτι ή αν και αυτό έχει ξεχαστεί. Ευχαριστώ. Julie Gerling. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Τίμερμανς. Σίγουρα συμφωνώ με τις προτεραιότητές σας ε, για το περιορισμό της γραφειοκρατίας ε, και για την καλύτερη νομοθεσία. Γι' αυτό κάπως μπερδεύομαι όταν ε, δεν μπορείτε να είστε ξεκάθαρος για τα θέματα του επικεφαλής Οικονομικού Συμβούλου. Όταν ερωτηθήκατε για τον επικεφαλής Οικονομικό Σύμβουλο, απαντήσατε ότι δεν ήταν, τέλος δεν ήταν ξεκάθαρη η απάντησή σας. Θα ήθελα λοιπόν να μας απαντήσετε τώρα γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση και τι είναι αυτό το οποίο δεν συμβαίνει. Κυρία Μιούλα, κύριε την Πρόεδρε, εδώ στην Επιτροπή μας συζητάμε ήδη τις προτάσεις Επιτροπής για την κλωνοποίηση και για την ε, γεωργία τι δυσκολίες υπάρχουν ε, ε, και σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις ε, στο πλαίσιο του TTIP. Και δεύτερη ερώτηση, το στρατηγικό πλαίσιο για την Ενεργειακή Ένωση. Μετά το 2020 πώς θα εφαρμόζεται το εμπόριο εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος και κατά πόσο επηρεάζεται η επίτευξη των στόχων για το 2020. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Président, merci. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε θα είμαι πολύ σύντομος. Σας ευχαριστώ πολύ για τα εισαγωγικά σας λόγια. Ε, γιατί είπατε πολύ σωστά ότι η ε, ανάπτυξη θα πρέπει να είναι κάτι το εγκάρσιο αλλά ε, η αηφόρος ανάπτυξη σημαίνει ότι θα πρέπει κανείς να βασιστεί στο δίκαιο και αυτό συνεπάγεται κάποιους κανόνες προστασίας. Επομένως ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα για την επίτευξη νέου δικαίου ε, σε μια γενικότερη κατάσταση παρακμής. Το δεύτερο ζήτημα μου αφορά την βιοπικιλότητα. Ε, μας δώσατε κάποια πληροφόρηση γι' αυτό, αλλά σήμερα αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση η οποία απαιτεί να αντιμετωπίσουμε το θέμα της βιοπικιλότητας όπως και το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Βρισκόμαστε στην, ε, στο έκτο κύμα ε, εξαφάνισης ειδών από δημιουργία της γης. Ε, σε λίγο θα φτάσουμε στα προβλήματα των ωκεανών. Ανοίγεται λοιπόν ένα νέο πεδίο και για την ανάπτυξη και για την έρευνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να παραμείνει ε, ηγέτιδα δύναμη μόνο εάν μαζικά επενδύσει στην θαλάσσια οικονομία. Και να μην λησμονούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πρώτη θαλάσσια δύναμη στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος αλλά όχι Ελλάσσον ο κύριος Μπλέμελης. Ευχαριστώ. Σε 9 μήνε ε, θα γίνουν ε, οι συζητήσεις οι μεγάλε ε, για την κλιματική αλλαγή στο Παρίσι και παραμένουν τα προβλήματα όσοι έχουν. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να επιτύχει ανάπτυξη εις βάρος του περιβάλλοντος, αυτό θα είναι μια πύρια νίκη σίγουρα. Ο Φράνσις Μπέικον είχε πει ότι εάν θέλουμε ε, αποτελέσματα χωρίς ε, που δεν τα έχουμε επιτύχει ποτέ θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουμε και πρωτόγνωρες μεθόδους. Νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε καινοτόμα ε, και μήπως θα μπορούσατε να μας διαφωτίσετε ποια θα μπορούσε να είναι η καινοτόμα σκέψη και δράση. <laughs> thank you for all those questions. I'm not sure. Ευχαριστώ για όλες αυτές τις ερωτήσεις. Δεν νομίζω ότι έχω αρκετό χρόνο, τόσο χρόνο όσο αξίζουν και δικαιούνται ε, για να τις απαντήσω. Ε, ο κ. Μπελέτ έχει δίκιο. Υφίσταται ένα σοβαρό πρόβλημα διαρροής υλικών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα δεν έχουν όλα τα κρατημένη το ίδιο νομικό πλαίσιο για να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο. Μιλούσα για παράδειγμα με Γάλλους επιχειρηματίες ε, ε, στον τομέα της, ε, του σκραπ στην Γαλλία. Όλες οι συναλλαγές θα πρέπει να, γίνουν, πρέπει να γίνονται με μέσα που δεν είναι μετρητά, δηλαδή επιταγές κλπ. Αυτό όμως δεν εφαρμόζεται σε χώρες όπως το Βέλγιο, η Γερμανία, οι κάτω χώρες κλπ. Όπου μπορούν οι πληρωμές να γίνονται με μετρητά. Πληρωμές με μετρητά σημαίνουν ότι γίνεται πολύ πιο δύσκολο να κλείσουμε όλα τα παραθυράκια. Γιατί γνωρίζουμε πώς λειτουργεί η αγορά του σκραπ. Ε, δεν είναι παράνομο λοιπόν. Το προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αλλά η διαφορά των εθνικών νομοθεσιών δημιουργεί συχνά τέτοιου παραθυράκια. Μιλώντας με τους επιχειρηματίες, μιλώντας με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανακαλύπτω και εγώ αυτά, αυτά τα κενά και σκέφτομαι μήπως θα έπρεπε να κάνουμε εμείς κάτι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ε, αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Σας λέω λοιπόν ότι το σκεφτόμαστε. Σε ό,τι αφορά τα φρούτα στα σχολεία, είναι αγαπημένο μου, προσφυλές μου θέμα. Η Κομισιόν εξετάζει το ζήτημα. Εγώ με τον Επίτροπο Χόγκαν ε, το εξετάζουμε. Η κατάσταση δεν συνάδει με την έκθεση του, ε, του συνεδρίου. Υπάρχει θέμα επικουρικότητας, σαφέστατα, αλλά το εξετάζουμε στην Κομισιόν. Για να ευθυγραμμιστούμε με το ελεκτικό συνέδριο, θα πρέπει να αναλάβουμε δράση αλλά δεν ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως καθήκον να αποφασίσει την παροχή φρούτων ή γάλατος στα σχολεία. Γνωρίζουμε τις απόψεις και τις λαμβάνουμε υπόψη πάντως. Και εγώ και ο κ. Χόγκαν. Για το θέμα της λογικής ε, συνέπειας και συνεκτικότητας, α, και ο κ. και επίσης έφυγε, οπότε αυτό με βοηθάει, θα τελειώσουμε και πιο γρήγορα. Για το θέμα της άγριας ε, πανίδας και τα εγκλήματα εναντίον της. Θα πρέπει να σας απαντήσω γραπτός γιατί ε, δεν είμαι ενημερωμένος αυτή τη στιγμή. Το ISDS, ο Μηχανισμός Επίλυσης Διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών στο πλαίσιο της TTIP. Ε, γνωρίζω τις ευθύνες μου, ευχαριστώ που μου το επιθυμίζετε, θα το εξετάσω στο τέλος των διαπραγματεύσεων. Όπως γνωρίζετε, η Κομισιόν εξετάζει διάφορες εναλλακτικές λύσεις αυτή τη στιγμή Θα αναλύσουμε και θα συζητήσουμε σε βάθος αν είναι απαραίτητο αυτός ο μηχανισμός και πώς θα εφαρμοστεί. Κατανοώ ορισμένες από τις ανησυχίες, από τους διθαγμούς, από τις εφυλάξεις. Κάποιοι βέβαια υπερβάλλουν λέγοντας ότι αυτός ο μηχανισμός θα σηματοδοτήσει το τέλος της δημοκρατίας. Υπάρχουν εκατοντάδες παρόμοιοι μηχανισμοί σε όλο τον κόσμο. Ίσως δεν είναι η τέλεια λύση, ίσως θα έπρεπε να διαθέτουμε ένα διεθνέ δικαστήριο, πλην όμως αυτό δεν θα δημιουργηθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Πάντως θα εξετάσουμε όλα τα επιχειρήματα. Νομίζω ότι και εσείς και πολλοί άλλοι έχουν ήδη βγάλουν συμπέρασμα. Οπότε αυτό είναι λίγο αντιφατικό. Μα ζητούν συχνά να εξετάσουμε κάτι πολύ προσεκτικά αυτοί οι οποίοι έχουν ήδη πάρει τι αποφάσει του και δεν έχουν σκοπό να κοιτάξουν το θέμα εξίσου προσεκτικά. Εν πάση περιπτώσει εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη να ε, δούμε το ζήτημα. Σίγουρα χρειάζεται να βελτιώσουμε την εφαρμογή της ε, νομοθεσία νομοθεσίας και ενδεχομένως να προσφέρουμε πιο πολύ ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εναντίον των παραβατών. Όμως αυτό δεν αφορά μόνο το περιβάλλον, αλλά και πολλούς άλλους τομείς. Πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Θέλουμε όλες οι δράσεις μας να είναι σύμφωνες με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής ε, Κομισιόν ε, και με τις αρχές της βελτίωσης νομοθεσίας. Δεν μπορώ να προδικάσω ε, τις ε, πρωτοβουλίες μας για το χρόνο εργασίας. σε ό,τι διαφορά την βιοποικιλότητα θα σας υποβάλω γραπτή την απάντησή μου ε, θίγει και στον πρώτο γύρο ερωτήσεων για να αποφύγουμε παρεξήγηση το πακέτο για την ποιότητα του αέρα δεν αποσύρθηκε εξακολουθεί να ε, είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων εξετάζουμε την τροποποίηση του μετά την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου αυτό είπα και στις άλλες επιτροπές και στους ε, εισηγητές Ο κ. Φλόρεντς με ρώτησε τι κάνουμε τώρα. Να σας πω το εξής. Θέλω κάθε φορά που βάλουμε προτάσεις για παράδειγμα για την κυκλική οικονομία να τηρούν τις ε, δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει και να ε, βρίσκονται να έχουν την ποιότητα την οποία έχουμε υποσχεθεί. Δεν πρόκειται να ε, προανακοινώνουμε ένα-δύο στοιχεία των ε, προτάσεών μας κρατώντας τις υπόλοιπες κρυφές. Όχι. όταν είναι έτοιμη η πρότασή μας θα την ανακοινώσουμε στο σύνολό της. Σε ό,τι αφορά το Μητρό Διαφάνειας θέλουμε να συμφωνήσουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υποχρεωτική ε, εγγραφή των ε, επαφών και συναντήσεων η Κομισιόν έκανε ένα πρώτο βήμα πολύ καλό δεν είναι το τέλος της ε, συζήτησης αυτό καλώς ορίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που κινείται προς την ίδια κατεύθυνση το ίδιο θα ήθελα να κάνουν και οι ίδιοι βουλευτές δηλαδή ή ε, τα άτομα τα οποία συναντώνται μαζί τους να, έχουν, να είναι υποχρεωμένα να εγγραφούν σε ένα κατάλογο. Νομίζω ότι από κοινού μπορούμε να εξετάσουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Και όλοι ε, θα βγούμε κερδισμένοι και οι τα δύο όργανα στη συζητήση με το Συμβούλιο να συμφωνήσουμε μεταξύ μας. Τώρα, για το θέμα της οδηγίας για το Habitat, ε, για Ε, τα οικοσυστήματα ε, δεν είμαι υπέρ της ε, μείωσης των του χαμηλώματος των προδιαγραφών στις κάτω χώρες πολλά προβλήματα δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο της οδηγίας πολλοί βέβαια το αρνούνται πολλοί υπουργοί γεωργίας το αρνούνται στις κάτω χώρες αυτό Εξακολουθώ να πιστεύω όμως ότι αν δείτε τη διαφορά στην μεταγραφή της οδηγίας μεταξύ των κρατών μελών ε, καταλαβαίνετε, θα καταλάβετε γιατί σε άλλες χώρες δημιουργήθηκαν προβλήματα και σε άλλες όχι. Επίσης μπορώ να επιβεβαιώσω ότι για τα θέματα των αποβλήποντων ε, είμαστε πολύ φιλόδοξοι. Το θέμα της ε, κυκλικής οικονομίας, όπως σας είπα, θα έχετε την πρότασή μέχρι το τέλος του χρόνου. θέλουμε να είναι έτοιμη έτσι ώστε να συμπέσει με την αρχή των σχεδίων του προγράμματος Juncker. Και από την κοινωνία και από τη βιομηχανία παίρνω θετικά μηνύματα. Ορισμένα από τα σχέδια ε, που θα εμπίπτουν στην χρηματοδότηση από ΣΔΙΤ είμαι σίγουρος ότι θα ε, εμπίπτουν, θα έχουν σχέση με αυτό ακριβώς στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Κύριος Ντάνκαν, ε, Σχολεί στο θέμα των εξετρών εξεδρών εξόριξης πετρελαίου στη θάλασσα και στην ε, Επιτροπή Βιομηχανίας ήδη απάντησα δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε κάποια διάκριση υπέρ τους. Θα το εξετάσω, βέβαια. Έχω την εντύπωση όμως ότι αν εύκολα πούμε ότι αυτές οι εξέδρες είναι διαφορετικές από όλα τα υπόλοιπα, ενδεχομένως οι εγκαταστάσεις καύσης θα μετακινηθούν προς τα εκεί, στη θάλασσα. Και αυτό βέβαια δεν θα ήταν υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης. Πάντως ε, θα του δώσουμε γραπτή απάντηση κ. Ντάνκαν. Σε ό,τι φορά τα φάρμακα, δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση αυτή τη στιγμή. Θα σας τη στείλω γραπτός, δεν ήμουν έτοιμος να μιλήσω για θέματα φαρμάκων και τιμής φαρμάκων σήμερα. Λυπάμαι. Θα σας στείλω απάντηση γραπτός. Τώρα, η κυκλική οικονομία είναι σημαντική για την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης. Ε, το ε, σχέδιο Juncker ε, το λαμβάνει υπόψη. Ασφαλώς υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχουμε αντιφατικές θέσεις, αντιφατικά νομοθετικά κείμενα. Ακόμα και εδώ μέσα στο Κοινοβούλιο η Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει διαφορετική άποψη σε ορισμένα θέματα από την Επιτροπή Γεωργίας. Όλα αυτά αποτελούν τμήμα της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος και της ποικιλία ε, ε, ε, πολιτικών απόψεων που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα υπάρχει ένα θέμα συνέπειας μεταξύ των νομικών κειμένων και έχουμε πολύ δρόμο να διατρέξουμε, όμως σε κάθε δημοκρατική κοινωνία προφανώς η κοινωνία θα πρέπει να βρίσκει ένα τρόπο ισορροπίας ανάμεσα στις διαφορετικές απόψεις Και προφανώς και εδώ πέρα στο, στο Κοινοβούλιο κάθε επιτροπή βλέπει την ισορροπία με διαφορετικό τρόπο. Σε ό,τι αφορά το θέμα της νομοθεσίας. Η οδηγία, όπως λέω, ε, είναι δεσμευτική σε ό,τι αφορά τους στόχους, αλλά επιτρέπει στα κράτη-μέλη να επιλέξουν το δικό τους τρόπο και τις δικές τους μεθόδους για την εφαρμογή της. Αυτή είναι η ουσία του ορισμού της ε, οδηγίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι χαλαρή. Αν θέλουμε ένα ενιαίο τρόπο στην εφαρμογή της νομοθεσίας, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε την οδηγία ως τρόπο νομοθέτησης. Χρησιμοποιούμε τον κανονισμό. Ο κανονισμός δεν χρειάζεται μεταγραφή. Αλλά σίγουρα οι οδηγίες δεν είναι χαλαρές. Τώρα, ποιου στόχου θα εγκαταλείψουμε. Κανένα στόχο δεν πρόκειται να εγκαταλείψουμε. Διατηρούμε την, το επίπεδο τη φιλοδοξία μα για την Ατζέντα 2020, του στόχου για τη βιώσιμη ανάπτυξη κλπ. κλπ. Αλλά σίγουρα η επίτευξη των στόχων αυτών σε διεθνέ επίπεδο δεν θα είναι εύκολη. Οι προτάσεις μα για την περίοδο μετά το 2015 βασίστηκε στις ε, εθνικές και διεθνεί μα δεσμεύσεις και θα σας θα υποβάλουμε έκθεση για το πόσο κοντά είμαστε σε αυτού του στόχου. Γιατί είναι εύκολο να θέτουμε στόχους, αλλά πρέπει να βλέπουμε και το πόσο πλησιάζουμε σε αυτούς. Σε ό,τι αφορά την κλωνοποίηση, δεν είναι ένα θέμα το οποίο γνωρίζω πολύ καλά, θα επανέλθω και για το θέμα των στόχων του 2020 απάντησα, βιοπικιλία επίσης αναφέρθηκα σε αυτήν, θα υποβάλουμε γραπτή απάντηση. Τέλος, να επαναλάβω το εξής, θέλω να συνεχίσουμε το διάλογό μας. Θέλω να συνεχίσουμε να συζητάμε, είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. και καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να σπάσουμε τα στεγανά όχι μόνο στην Κομισιόν αλλά και στο Ευρωπαϊκό Ένα κόμμα σε ένα κράτος μέλος επιθυμεί να ξέρει τα πάντα για το πώς παίρνουμε επιστημονικές συμβουλές. Με ρώτησαν κάποια στιγμή αν ο πρόεδρος ε, της Κομισιόν θα κάνει αυτό που υποσχέθηκε στην ομάδα μας. Ναι, η απάντηση είναι ναι. Ο πρόεδρος της Κομισιόν θα κάνει αυτό που υποσχέθηκε σε αυτή την ομάδα και θα φροντίσει με σε στενή συνεργασία με τον ότι η Κομισιόν θα διαθέτει την πιο κατάλληλη και την καλύτερη δυνατή ε, επιστημονική ε, συμβουλευτική που μπορεί να εξασφαλίσει. Θα σας ενημερώσω μόλις η Κομισιόν αποφασίσει πώς θα γίνει αυτό. Grazie Vicepresidente Timmerman, eh, un sincero ringraziamento penso a nome di tutti i componenti della... Ευχαριστούμε τον Πρόεδρο Τίμερμαντ και νομίζω ότι εκ μέρους όλων των μελών της Επιτροπής μπορούμε να σας ευχαριστήσουμε όχι μόνο γιατί μας δώσατε που μας περισσότερο χρόνο για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις αλλά και γιατί θα λύσατε να δώσετε λεπτομεριώς τις απαντήσεις στους περισσότερους συναδέλφους απαντώντας μεμονωμένα σε όλες τις ερωτήσεις που ετέθησαν. Διακόπτουμε για λίγο για να μπορέσει ο Αντιπρόεδρος να αποχωρήσει. Εμείς θα συνεχίσουμε τις εργασίες της Επιτροπής γιατί παραμένουν σημεία στην ημερησία Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος τώρα της, της συνεδρίασής μας. Ε, στις ε, ανακοινώσεις ε, του Προέδρου είναι το τρίτο σημείο. Μια διακοινοβουλευτική επιτροπή για τα θέματα της COP 21 για την ε, οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος θα γίνει στις 33 ε, το απόγευμα της Δευτέρας και θα ακολουθήσει και μία δεξίωση. Σας παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε αυτή την ε, συνάντηση με τα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ε, νομίζω ότι τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίας μπορούν να θεωρηθούν ότι εγκρίνονται. Για το σημείο 5 θέλω να ενημερώσω τα μέλη της Επιτροπής για τον τριμερή διάλογο για τα νέα τρόφιμα. Στον τρίτο διάλογο που έγινε στις 26 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τη στρατηγική που ορίστηκε στα έγγραφα της συνεδρίασης, παραμένει ένα ε, σημαντικό πολιτικό θέμα το θέμα ε, συζητήθηκε η κλωνοποίηση, τα ανανοηλικά, η κατεξουσιοδότηση πράκτης, η αρχή της προφύλαξης ε, και παρότι ε, καταλήξαμε σε μια καταρχήν συμφωνία για τα περισσότερα πολιτικά θέματα, χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση για τα θέματα της κλωνοποίησης και για την δέσμη μέτρων για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Χρειάζονται και άλλα βήματα για να μπορέσει να γίνει ο επόμενος τριμερής διάλογος που έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Μαρτίου, ούτως ώστε να καταλήξουμε σε μια τελική πολιτική απόφαση. Και τώρα πρέπει να συζητήσουμε στο σημείο 6 την γνωμοδότηση για την πράσινη οικονομία και θα δώσω κατευθείαν το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Εύη. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα σας κάνω μία πρώτη εισαγωγή για να σας πω ότι η δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας δεν μπορεί να θεωρηθεί απλώς στόχος αλλά σαν ε, θετικό παράλληλο επίτευγμα ε, στα πλαίσια της ικανοποίησης των δικών μας ε, απαιτήσεων για την περιβαλλοντική αηφορία θέλουμε να δημιουργήσουμε τις οικονομικές περιβαλλοντικές προϋποθέσεις που θα έχουν σαφείς στόχους, φιλόδοξες ε, ε, αρχές καθώς επίσης και την δυνατότητα να προωθήσουν ακριβώς την πιο ε, πράσινη οικονομία. Στο Ευρωβαρόμετρο ε, αναφέρεται ότι αυτές οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι πιο πράσινες μπορεί να έχουν πάρα πολύ καλά κλιματικά αποτελέσματα όσον αφορά ας πούμε την εξοικονόμηση ενέργειας. Επίσης ε, θα πρέπει να προχωρήσουμε μέσα από δεσμευτικούς νομοθετικούς κανόνες οπωσδήποτε σε ενωσιακό επίπεδο και να δημιουργήσουμε δημιουργήσουμε τις ε, θετικές προϋποθέσεις ε, για την ολοκλήρωση της κυκλικής οικονομίας ε, όπου τα υλικά της ανακύκλωσης θα χρησιμοποιούνται σαν πρώτα και δεύτερα υλικά. Θα πρέπει οπωσδήποτε πρώτα απ' όλα να ταυτοποιήσουμε αυτά τα οικονομικά και επιχειρησιακά εργαλεία τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να επιτύχουμε τους στόχους μας. Σκεφτήκαμε ότι και εδώ ο καθορισμός δεσμευτικών στόχων, στόχων αφορά την ε, οικονομική, ε, συγγνώμη, την ενεργειακή ε, εξοικονόμηση κτλ. θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα εργαλείο εξαιρετικά χρήσιμο για τις υπηρεσίες εκείνες οι οποίες δεν έχουν την δυνατότητα από μόνες τους, κυρίως τοπικές αρχές που δεν έχουν την δυνατότητα από μόνες τους να πάρουν μέτρα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να τεθούν δεσμευτικοί στόχοι όσον αφορά τον χρήση, τον, τις χρήσεις ανανεώσιμων πόρων και της εξοικονόμησης ενέργειας, φωτοβολταϊκά πάνελ κτλ. Επίσης ε, σε τομείς οι οποίοι δεν καλύπτονται από το EDS ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφερθούν στόχοι συγκεκριμένοι όσον αφορά την εκπομπή ρήπων. Θα πρέπει οπωσδήποτε η ανάπτυξη να γίνεται μέσα από πράσινες υπηρεσίες ε, και οι επαγγελματίες θα πρέπει να έχουν κυρίως στον οικοδομικό τομέα και κατάρτιση όσον αφορά τα, ε, τις ε, πιο πράσινες ε, επιλογές που μπορούν να κάνουν. Για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τον στόχο μας όσον αφορά τα απόβλητα θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να ληφθούν συγκεκριμένα δεσμευτικά μέτρα. Ε, η ανακύκλωση των υλικών και η ε, επιλεκτική συλλογή αποβλήτων και απορριμμάτων θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη οι οποίες μπορούν και πρέπει να ακολουθηθούν από όλους. Θα πρέπει επίσης ε, να δοθούν κίνητρα έτσι ώστε από την αρχή ε, της διαδικασίας, δηλαδή από την έρευνα μέχρι το τέλος που είναι η βιομηχανική εφαρμογή, να δίνονται λέω τα απαραίτητα κίνητρα έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε και τις μολυντικές διεργασίες αλλά και να μειώσουμε το κόστος το οποίο τελικά πληρώνει ο καταναλωτής. Θα πρέπει να δημιουργηθούν πράσινες θέσεις εργασίας αλλά πριν γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Εναρμόνιση λοιπόν σε ευρωπαϊκό ε, ενωσιακό επίπεδο όσον αφορά την φορολόγηση η οποία από τη φορολόγηση εργασίας ε, θα πάει στη φορολόγηση της ε, κατανάλωσης. Μια τέτοια υπόθεση εργασίας οπωσδήποτε θα έκανε πιο αποτελεσματική τη χρήση ε, της ε, σήμανσης ε, eco-label και θα μπορούσε επίσης να έχει αντίκτυπο και στην GPP, αυτή δηλαδή την διαδικασία για τους πράσινους δημόσιους διαγωνισμούς. Κατά αυτή την έννοια πιο πράσινα προγράμματα θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη επιτυχία στους ε, πράσινους, να ωφελούνται περισσότερο σε αυτούς τους πράσινους δημόσιους διαγωνισμούς. Επίσης ε, θα πρέπει να θυμίσουμε και κάποια αριθμητικά στοιχεία. Υπάρχουν συγκεκριμένες μελέτες ε, οι οποίες αναφέρουν ότι ένα δις δαπάνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ε, την ε, ε, ενεργειακή ανασύνθεση και που μπορούν να δημιουργήσουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Ενώ εάν το ίδιο δις χρησιμοποιηθεί με παραδοσιακούς τρόπους θα έχει οπωσδήποτε πολύ μικρότερο αντίκτυπο όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Να πούμε επίσης ότι υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια έτσι ώστε να δημιουργηθούν πράσινες θέσεις εργασίας οι οποίες άμεσα μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσα από την ενεργοποίηση ακριβώς αυτών των βελτίστων πρακτικών που ήδη υφίστανται και μέσα από την προώθηση καινοτόμων ερευνητικών και βιομηχανικών διεργασιών. Σήμερα μας τα είπε άλλωστε και ο Αντιπρόεδρος Τίντερμανς ότι εάν δεν ε, ότι εφόσον τα κράτη-μέλη δεν ε, ε, εφαρμόζουν την υφιστάμενη νομοθεσία, οπωσδήποτε επιβραδύνεται το πρασίνισμα της... Δεν είναι δυνατόν να λησμονήσουμε ότι ε, υπάρχει και αυτό το πρόβλημα με τη δέσμη για τα απόβλητα ε, που έχει αποκλείσει τη δημιουργία τουλάχιστον 400.000 θέσεων πράσινης απασχόλησης. Αυτά ήθελα να σας πω σε μία πρώτη φάση και είμαι βεβαίως στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ σας, ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Μπορούμε τώρα να δώσουμε το λόγο στους ε, σκιώδεις εισηγητές. Ο κύριος Ανδρουλάκης παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το πολύ καλό σχέδιο γνωμοδότησης που προετοίμασα. Είναι μια πολύ καλή βάση η οποία μπορεί να συμπληρωθεί από κάποια επιπλέον στοιχεία. Παρά την κακώ εδρεωμένη άποψη ότι η πράσινη οικονομία αφαιρεί θέσει εργασία, οι δυνατότητε απασχόληση που δίνονται είναι πολλέ και σε μεγάλο βαθμό αναξιοποιητέ. Έχει παρατηρηθεί ότι οι πράσινε θέσει εργασία είναι πιο ανθεκτικέ στου οικονομικού κύκλου. Είναι λοιπόν προ το συμφέρον μα να επιδιώξουμε την περαιτέρω ανάπτυξη τη πράσινη οικονομία. Υπολογίζεται πω αν εφαρμοζόταν πλήρω η υπάρχουσα νομοθεσία για τα απόλυτα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μερικέ χιλιάδε νέε θέσει εργασία σε όλη την Ευρώπη. Και όπω αναφέρθηκε στην νομοδότηση, η απόσυρση τη πρόταση για την αναθεώρηση των οδηγιών αυτών υπονομεύει τη δημιουργία επιπλέον 180.000 θέσεων εργασία. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο να φέρουμε την ανάγκη άμεση υποβολή καινούργια πρόταση, αλλά να επισημάνουμε και εκείνα τα σημεία τα οποία είναι απαραίτητα και τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση τη απασχόληση, όπω ανέφερε και η προηγούμενη συγγήτρια. Στο ίδιο πλαίσιο, η νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και η εφαρμογή τη οποία θα μπορούσε να συνεισφέρει στη μείωση τη ανεργία και σε ένα κλάδο όπω ο κατασκευαστικό, που πλήγεται ιδιαίτερα στι χώρε που περνούν κρίση, όπω η δικιά μα χώρα για την περαιτέρω ανάπτυξη τη πράσινη οικονομία αλλά και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνονται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασία, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, σε περιβαλλονομένου βεβαίω και του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Συγχρόνω, θα πρέπει να έχουμε το μυαλό μα και στην ομαλή μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών ρήπων, χωρί όμω να θέτουμε σε κίνδυνο θέσει εργασία που κινδυνεύουν από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Για το λόγο αυτό, με τροπολογία μα ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άμεση αναθεώρηση του συστήματο εμπορία δικαιωμάτων ρήπων, διατηρώντα όμω ένα σύστημα προστασία για τι βιομηχανίε που πλήττονται από το carbon leakage και μετά το 2020. Τέλο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο θέμα τη περιβαλλοντικής φορολογία, η οποία δεν θα πρέπει να επιβαρύνει τον απλό καταναλωτή. Ολοκληρώνοντα, θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι την συγκήτρια για το πολύ καλό σχέδιο γνωμοδότηση που ετοίμασε και ευελπιστώ σε μια καλή συνεργασία μαζί της καθώς και με τους υπόλοιπους πιο δεσηγητές. Thank you very much. And now, Mr. Duncan. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντάνκαν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η ομάδα του ECR χαιρετίζει σε γενικές γραμμές ε, την πρόταση αυτή. Υπάρχουν πολλά ε, θετικά στοιχεία, θα κάνουμε κάποιες ε, προτάσεις. Πιστεύω ότι δεν τονίζεται η πρόοδος που έχει ήδη γίνει σε πολλούς τομείς που ήδη έχουν κάνει πολλές προσπάθειες, Παραδείγματο χάρη αυτοκίνητο βιομηχανία, χημική βιομηχανία κλπ. Και είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε αυτά τα οποία ήδη έχουν γίνει και θα αποτελέσουν μια πλατφόρμα για αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν και για να υπάρξει μια κοινή πλατφόρμα βέλτιστων πρακτικών. θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και τις προκλήσεις ε, που υπάρχουν ε, και για τη ε, διαρροή άνθρακα. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχουν και κίνδυνοι και αν δεν προσέξουμε ιδιαίτερα θα υπάρξουν πολλές συνέπειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, πολύ κίνδυνοι για τη βιομηχανία γενικότερα. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε κάποιου από αυτού του βασικού κινδύνου όταν μιλάμε για τι πρωτοβουλίε αυτέ. Τώρα, συγκεκριμένοι κίνδυνοι, ε, συγκεκριμένε ανησυχίε. Ε, η φορολογική πολιτική δεν είναι αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένει αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και όταν η έκτη παράγραφο μιλά για αναρμόνιση φόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε, διότι δεν είναι αντικείμενο αυτής της πρωτοβουλίας. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν ευελιξία για να μπορούν να σχεδιάζουν τη δική τους προσέγγιση σε, στα θέματα βιομηχανίας χαμηλού άνθρακα και υψηλής απασχόλησης και όχι να καταφεύγουμε στον χαμηλότερο κοινό παρονομαστή. Θα πρέπει από την τωρινή κατάσταση που ε, σε γενικές γραμμές ε, είναι οι βιομηχανίες ε, με τα βάρη του παρελθόντος θα πρέπει να περάσουμε ε, στη μελλοντική κατάσταση που θα μπορέσουμε να κάνουμε σημαντικές συνεισφορές για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βέντε. Χωρίς μικρόφωνο. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεσή της ε, που τονίζει τη σημασία δημιουργία πράσινων θέσεων απασχόληση. Ε, πολλά μέτρα πρέπει να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κατών μελών για να ενισχύσουμε την πράσινη απασχόληση. Θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ε, πράσινες θέσεις απασχόλησης όπως λέει η εισηγήτρια σε διάφορα σημεία και συμφωνώ μαζί της πρέπει να θέσουμε στόχους ενεργειακής αποδοτικότητας και γι' αυτό η Επιτροπή πρέπει το συντομότερο δυνατόν να μας υποβάλει φιλόδοξες προτάσεις. Παρότι οι προτάσεις αυτές είναι σημαντικές, δεν είναι επαρκείς. Σύμφωνα με την, τον Ευρωπαϊκό Φορέα Περιβάλλοντος, την έκθεση του την προηγούμενη εβδομάδα, χρειάζεται περισσότερα μέτρα η Ευρώπη για να επιτύχει του στόχου του 2050. Πρέπει να πλησιάσουμε πιο γρήγορα μια ε, πράσινη οικονομία θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μέχρι και ένα εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας στον τομέα των μεταφορών αν έχουμε αυστηρά μέτρα όσον αφορά τον, τις εκπομπές και προωθήσουμε τις ε, ηλεκτρικές μεταφορές. Η μόνωση κατοικιών και η θέρμανση επίσης είναι τομείς που θα μπορέσουν να βοηθήσουν ε, την πράσινη ε, ανάπτυξη και αν έχουμε και τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία. Επίση, θα δημιουργηθούν νέε θέσει απασχόληση. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το πρόγραμμα επενδύσεων του Προέδρου Juncker που θα προσφέρει 315 δισεκατομμύρια στην ε, οικονομία τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να φροντίσουμε να συνεισφέρει στην πράσινη οικονομία και ιδιαίτερα θα πρέπει να τονίσουμε ότι θα πρέπει η έρευνα και η καινοτομία να είναι βασικά συστατικά οποιοδήποτε μέτρου στην κατεύθυνση της Ευρώπης του 2020. Θέλουμε όχι μόνο θέσεις απασχόλησης, αλλά ε, βιώσιμες πράσινες θέσεις απασχόλησης. Ελπίζουμε ότι μέχρι το 2020 ακόμη και 1,5 εκατομμύριο θέσεις απασχόλησης μπορούν να δημιουργηθούν αν οι κυβερνήσεις χειριστούν καλύτερα το σύστημα εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για άλλη μια φορά και προσβλέπω στη συνεργασία μαζί της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω. την για τη δουλειά τη. Ε, είναι αργά ήδη, κάποιοι άλλοι συνάδελφοι ήδη είπαν αυτά που είχαν να πω. Δεν θέλω να, ε, να κρηγορήσω. Θα πρέπει απλώς να αντιληφθούμε ότι το ότι βάζουμε κάτι σε ένα χαρτί εδώ στη Βρυξέλλες αυτό δεν σημαίνει ότι θα εφαρμοστεί στα κράτη-μέλη. Μ' αρέσει αυτό που λέγεται, ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν την ευθύνη ε, και να κάνουν δικό τους όλο αυτό το ε, πρόγραμμα. Δεν πρέπει απλώς ε, να έχουμε κοινέ αρχές, ε, θα πρέπει να, τα κράτη-μέλη να είναι πολύ ενεργά και δραστήρια στην εφαρμογή των νομοθετικών κειμένων. Πιστεύω όμως ότι ε, θα πρέπει να δώσουμε και στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα αυτή με περισσότερες κατευθυντήριες γραμμές, για παράδειγμα, για τα χρονοδιαγράμματα κλπ. Το... Οι προτάσεις ε, Juncker δείχνουν ότι θα ε, χρηματοδοτήσουν τα πάντα. Τις ε, ε, πράσινες ε, θέσεις εργασίας, την Ενεργειακή Ένωση, τα πάντα. Όμως αυτή τη στιγμή το, οι προτάσεις Juncker είναι στο χαρτί ε, η χρηματοδότηση ε, θα βασιστεί στις αποφάσεις των κρατών μελών τελικά και των επιχειρηματιών. Εμείς θα πρέπει να διευκολύνουμε απλώς αυτή τη χρηματοδότηση. Οπότε θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η προσθέμενη αξία κάθε φορά των δράσεων. Με βάση αυτή την προστέμενη αξία θα διευκολύνουμε τη χρηματοδότηση προς, τη μία προς την άλλη κατεύθυνση. Θα πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε στενά με τα κράτη-μέλη και κάτι άλλο. για την παρέμβαση που επιχειρείται στα φορολογικά στήματα των κρατών μελών. Νομίζω ότι αυτό θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Τα κράτη-μέλη συνήθως δεν θέλουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Ε, αυτή τη στιγμή η διατύπωση όμως δεν είναι πολύ σαφής ε, και μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Χρειάζεται προσοχή για να μην υποσκάψουμε και τα υπόλοιπα που έχει το κείμενο και είναι θετικά. Ευχαριστώ. Οι πράσινε θέσει εργασία αποτελούν τμήμα μια ολόκληρη διαδικασία μετασχηματισμού κοινωνικού και οικονομικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, αποτελούν εγγύηση μια ε, βιώσιμη ανάπτυξη και βιώσιμη οικονομία. Καλωσορίζω την ε, έκθεση τη Ελεονόρα και θα ήθελα να κάνω τα εξής σχόλια. Θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία της ε, ε, κυκλικής οικονομίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τηρήσει τις υποσχέσεις της, να παρουσιάσει ένα πιο φιλόδοξο πακέτο μέτρων μέχρι το τέλος του χρόνου. Εξ, εξαρτώμεθα όλο και περισσότερο από τις ε, πρώτες και αυτές οι πρώτε ε, απειλούν την σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η σταθερότητα μπορεί να εξασφαλιστεί μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο θα περιλαμβάνει το συντονισμό των, ε, της ε, κανονιστικής ε, ρυθμιστικής και οικονομικής πολιτικής οι στόχοι θα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμοι και δεσμευτικοί έτσι ώστε πραγματικά να προωθήσουμε ε, τις ε, επενδύσεις ε, και την αποτελεσματική χρήση των πόρων και των κονδυλίων. Όλα αυτά θα οδηγήσουν σε μια μεταμόρφωση της ευρωπαϊκής οικονομίας που θα την καταστήσει πιο ανθεκτική έναντι των οικονομικών κύκλων. Οι πράσινε τέσσερα εργασία είναι σημείο κλειδί σε, σε αυτό το μετασχηματισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν η συνάδελφο Εύη θέλει να ξαναπάρει το λόγο. Ναι, μόνο ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα λόγια τους και να υπογραμμίσω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταφέρουμε να δώσουμε θετικά μηνύματα έτσι ώστε να συμβεί η αλλαγή ε, γιατί ε, εάν δεν γίνει αυτή η αλλαγή ή μάλλον να το θέσω διαφορετικά, εάν δεν καταλάβουμε όλοι και αν δεν συμβάλλουμε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση, ε, τότε δεν πρόκειται να φτάσει και το καλό αποτέλεσμα. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη επίσης και όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν για τα φορολογικά, για την ε, κυκλική οικονομία, γιατί διαφορετικά χωρίς αυτό η Ευρώπη δεν θα επιτύχει τους στόχους της. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και σίγουρα σύντομα θα τα ξαναπούμε, έτσι ώστε και με τη δική σας όθηση να βελτιώσουμε τα πράγματα. 17 Μαρτίου στις 12 λίγη η προθεσμία για τις τροπολογίες, 6-7 Μαΐου ψήφος στην ε, Επιτροπή μας, 28 Μαΐου στην Επιτροπή Απασχόλησης που είναι η αρμόδια καθήλη ε, και στην Ολομέλεια Ιούνιο ή Ιούλιο, δεν ξέρουμε ακόμα, δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν έχουμε κάτι στα διάφορα. Καλό σας βράδυ.